Guten Morgen. Morning, ladies and gentlemen. Καλημέρα, κυρίε και κύριοι. So on. Are you ready? Can we start? Μπορούμε να ξεκινήσουμε. Ja, Guten Morgen, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Καλημέρα, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Σας ε, καλωσορίζω στην πρώτη αυτή συνεδρίαση του νέου έτους. Επί τη ευκαιρία σας εύχομαι και ευτυχές υγιές ε, το 2012 και εύχομαι και ελπίζω να συνεχιστούν οι εργασίες μας ε, στην Επιτροπή. Έχουμε σημαντική δουλειά να συνεχίσουμε, νέα πράγματα να αρχίσουμε. Το 2012 λοιπόν προβλέπεται έτος ε, στο οποίο θα έχουμε τουλάχιστον την ίδια ε, δουλειά, αν όχι και περισσότερη. Όσον αφορά τις παρατηρήσεις του Προέδρου, στα σημεία 1 και 2, πρώτα απ' όλα για την ημερήσια διάταξη άλλαξε η σειρά των σημείων. Το ξέρετε, νομίζω πως το σημείο 6 ε, πήγε μεταξύ 3 ε, και 4 εάν δεν υπάρχει κάποια αντίρρηση τότε εγκρίνεται η ημερήσια διάταξη όπως τροποποιήθηκε να σας ανακοινώσω επίσης κάποια πραγματάκια πρώτον ο κύριος Μπάιερ δίπλα μου ανέλαβε τα νέα του καθήκοντα ως επικεφαλής της μονάδας της γραμματείας της Επιτροπής μας. Τον καλωσορίζω, εύχομαι καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα και καλή δουλειά και καλά μυαλά. Και έτσι πλέον είναι ξεκάθαρα τα πράγματα όσον αφορά την διεύθυνση της γραμματείας μας και χαίρομαι. Επί τη ευκαιρία όμως, να ευχαριστήσω τον Ρίντζε Φαν Άρομ για την δουλειά του γιατί ήταν δύσκολα τα πράγματα. Τι έκανε. Έκανε τη δουλειά χωρίς να είναι υπεύθυνος ε, ούτε βεβαίως ε, ε, επισήμως την έκανε, αλλά ανέλαβε μια μεγάλη ευθύνη και έκανε εξαιρετικά αυτή τη δουλειά. Και θέλω να τον ευχαριστήσω εξ ονόματος όλων ημών. Σας ευχαριστούμε λοιπόν πάρα πολύ για τη δουλειά σας και την αξιοπιστία που επιδείξατε. Κατόπιν, να καλωσορίσω τον Ρούπερτ Βίλκινσον νέο μέλος της γραμματείας μας. Είναι εκεί στην τρίτη σειρά, τέρμα δεξιά. Καλώς ήρθατε στην Επιτροπή μας και καλή δουλειά εύχομαι τα επόμενα χρόνια και ταυτόχρονα να αποχαιρετήσω τον Siegfried Μπράιερ. Λοιπόν, ο οποίος μας εγκαταλείπει και βεβαίως είναι δύσκολο να αλλάζει κανείς ε, θέση. Τον ε, ευχαριστώ όμως, μας βοήθησε όλους και εμένα ε, προσωπικά, ειδικά όσον αφορά την προετοιμασία των συνεδριάσεων. Φρόντιζε να κύλουν τα πράγματα ομαλά. Σας ευχαριστούμε λοιπόν πάρα πολύ κύριε Μπράιερ. Ε, Κατόπιν να υπενθυμίσω πως η διοίκηση του Κοινοβουλίου είπε πως οι επιτροπές πρέπει να χρησιμοποιούν αποτελεσματικότερα το χρόνο μας για να εκμεταλλευόμαστε καλύτερα και τους πόρους της ε, διερμηνίας ότι δηλαδή θα πρέπει να συνεδριάζουμε Δευτέρα με Πέμπτη κανονικά, όχι μόνο τις ώρες και μέρες εχμής και από την άλλη ε, λέμε πως ε, θα πρέπει να ξανασκεφτούμε το να επικεντρωνόμαστε σε δύο μόνο μέρες. Γιατί βλέπετε ότι εμείς συχνά χρειαζόμαστε τρεις μέρες για να ολοκληρώσουμε τη δουλειά μας. Θα δούμε τώρα θα γίνει με το χρονοδιάγραμμά μας. Άλλη μια συζήτηση είχε γίνει με την Προεδρία της Δανίας, να το ξέρετε, όπου συζητήσαμε τους διάφορους ε, φακέλους. Ε, η Προεδρία ενδιαφέρεται να ολοκληρωθούν γρήγορα, αλλά και με τρόπο λογικό όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση βλέπετε πως ήταν ε, πολύ διαφορετική κατάσταση, αλλά δεν υπήρξε τίποτα το νέο, το γνωρίζουμε. Με την Ενίζα υπάρχουν δυσκολίες στο Συμβούλιο, αυτό το ξέρουν όλοι. Εγώ είπα πως εμείς τη δουλειά μας την κάναμε και πρέπει να προχωρήσουν ε, τα πράγματα από εκεί και πέρα. Δεν είναι τίποτα μικρολεπτομέρειες, είναι ένα κεντρικό πολιτικό ζήτημα και παραπονιόμαστε συνεχώς πως υπάρχει πρόβλημα, αλλά κανείς ε, δεν είναι διατεθειμένος να το λύσει. Ε, δεν είναι κατάσταση αυτή. Αυτά νομίζω αρκούν ε, ω εισαγωγή και περνάμε στο πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Έχουμε χρόνο μέχρι τις 10. Θα δούμε τώρα πώς θα κυλήσουν τα πράγματα. Είχαμε πει πως θα πρέπει να ξαναμιλήσουμε για την ενεργειακή απόδοση, γιατί θα πρέπει να μιλήσει κάποτε και η Κομισιόν που δεν μίλησε την προηγούμενη φορά γιατί είναι σημαντικό να ε, έχουμε μια ανοιχτή συζήτηση για αυτό το θέμα. Γι' αυτό η δική μου επιθυμία είναι να ξεκινήσουμε δίνοντας τον λόγο στην ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μετά να συζητήσουμε τα ανοιχτά ζητήματα. Καλά, ανοιχτά είναι πολλά, αλλά τα κύρια ζητήματα. Καλωσορίζω λοιπόν την κυρία Μαρίτα Ντόνελη και τις δίνω αμέσως τον λόγο. Σας ευνηδιάζω έτσι, αλλά σας είπανε φαντάζομαι τι συζητήσαμε την προηγούμενη φορά και θα ήθελα να σας παρακαλέσω να τοποθετηθείτε από πλευράς Κομισιόν για το θέμα το οποίο μας απασχολεί. Έχετε λοιπόν το λόγο. Κυρία Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ήθελα επί τη ευκαιρία να ευχηθώ καλή χρονιά σε όλους και επιτυχία μέσα σε αυτό το νέο έτος στο πλαίσιο της ενεργειακής απόδοσης. Είμαστε αισιόδοξοι ότι θα είναι επιτυχής η νέα χρονιά σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα. Η πρόταση ενεργειακής απόδοσης που αποτελεί μια από τις πρώτες προτεραιότητές μας βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη αυτή τη στιγμή. Χαίρομαι που βλέπω ότι η Επιτροπή και το Κοινοβουλίο προτιθένται να προχωρήσουν το ζήτημα όσο γίνεται πιο γρήγορα, το ίδιο και η Δανέζικη Προεδρία. Ελπίζουμε με ούριο άνεμο, ίσως και ε, ανανεώσιμο άνεμο, έτσι να καταλήξουμε σε καλά συμπεράσματα θα σας υποστηρίξουμε εμείς όσο γίνεται περισσότερο ώστε να επιτύχουμε όλους τους στόχους. Θα ήθελα να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία για να εστιαστώ σε τρία-τέσσερα ζητήματα κλειδιά της πρότασης. Το πρώτο που θα ήθελα ε, να αναφέρω αφορά τις ε, δημόσιες ε, συμβάσεις. Κάποιος την είπε ότι οι δημόσιες συμβάσεις έτσι όπως αναφέρονται στην πρόταση για την ενεργειακή απόδοση ίσως να μην συμμερφώνεται με την οδηγία για τις δημόσιες συμβάσεις του Δεκεμβρίου. Σας διαβεβαιώ ότι έχουμε συνεργαστεί στενά με τους συναδέλφους της εσωτερικής αγοράς πριν κάνουμε την πρόταση και υπάρχει απόλυτη συνοχή και συμμόρφωση. Η πρόταση δημοσίων συμβάσεων ε, λαμβάνει υπόψη και όλα αυτά εδώ είναι σημαντικό αυτό για την πρόθεση τη ενεργειακή απόδοση και των σχετικών εφαρμογών σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ένα δεύτερο βασικό στοιχείο της πρόταση είναι οι υποχρεώσει ενεργειακή απόδοσης. Η φιλοδοξία επίση που σχετίζεται με αυτές τις υποχρεώσεις. Έχουμε έναν βασικό στόχο και το επίπεδο φιλοδοξία που έχουμε συμπεριλάβει στην πρότασή μας το 1,5% είναι θεμελιώδες ε, παράγοντας ε, για να επιτύχουμε το στόχο. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν ενώ επικροτούμε την ενίσχυση ε, της επαλήθευσης και την αντιμετώπιση της έλλειψης καυσίμων θέλουμε να διατηρήσουμε το φιλόδοξο αυτό κείμενο. Ένα άλλο ζήτημα όσον αφορά την, ε, τις χρεώσεις και τη δημολόγηση. Αυτό αφορά άμεσα τους καταναλωτές. Οι καταναλωτές ε, μπορούν ε, να γνωρίζουν τι κάνουν μόνο εφόσον λαμβάνουν πληροφορίες και να λειτουργούν πιο ανεξάρτητα. Εδώ λαμβάνουν κάποιες πληροφορίες αλλά όχι επαρκείς. Γι' αυτό το λόγο ε, στην πρόταση ε, προτείνουμε να υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες προς του καταναλωτές ώστε να γνωρίζουν τι κάνουν, εξοικονομούν ενέργεια και να διαχειρίζονται την καταναλωσή τους. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό οι διατάξεις ε, μέτρησης και χρέωσης να υποστηρίζουν στο μέγιστο βαθμό τους καταναλωτές. Τέλος, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να απευθύνω ένα τελευταίο ζήτημα, το ζήτημα των στόχων είτε αυτή είναι δεσμευτική, είτε εθνική, είτε οτιδήποτε άλλο, είναι ένα σημαντικό σημείο και σε αυτό το πλαίσιο υποστηρίζουμε το Κοινοβούλιο σε οποιοδήποτε τεχνικό έργο που θα χρειαστεί να γίνει. Στο πλαίσιο της ανάλυσης υποστηρίζουμε επίσης το Συμβούλιο και ελπίζουμε ότι θα υπάρξει δυνατότητα να επιτύχουμε τον γενικότερο στόχο του 20% το αν αυτό θα το κάνουμε μέσω επιμέρου στόχων θα καθοριστεί ε, στη διαδικασία και κατά τις συζητήσεις μας. Αυτά είχα να πω τώρα κύριε Πρόεδρε. Καταλαβαίνω ότι έχουμε λίγο χρόνο. Ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε να μιλήσω και θα απαντήσω με ευχαρίστηση σε οποιασδήποτε ερωτήσει θέλετε μετά από τη συζήτηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάποιοι έχουν ε, ζητήσει τον λόγο. Ε, θα σας τον δώσουμε τη σειρά αν, δεν ζητήσει κάποιο άλλο. Ε, ναι. Λογικό ήταν να θέλει να μιλήσει και ο εισηγητή. Κλοντ, λοιπόν, έχει πρώτο λόγο. Τώρα δεν θέλω να βγάλω μεγάλους λόγους στην αρχή. Ε, θέλω απλά στο τέλος να μπορέσω να απαντήσω στου συναδέλφου. Τώρα, πληροφοριακά, γιατί δεν είναι για σας εύκολο να ξέρετε που είμαστε στη συνεδρίαση των Σκιωδών. Είχαμε δύο τέτοιες συνεδριάσεις και με βάση τη συζήτηση της προηγούμενης φοράς όπου κάποιοι συνάδελφοι είπαν είναι δυνατόν τέλος Ιανουαρίου να ψηφίσουμε ήδη ε, και ε, συζητήσαμε ανοιχτά για το πόσο γρήγορα μπορούμε να κινηθούμε και συμφωνήσαμε όλοι πως καλύτερα να ψηφίσουμε τέλος Φεβρουαρίου το οποίο θα μας επιτρέψει να έχουμε άλλες πέντε συνεδριάσεις των σκιωδών εισηγητών για να μπορέσουμε έτσι να έχουμε χρόνο να δούμε αυτές 1800 ε, τροπολογίες. Και Ε, Βεβαίω διαπραγματευόμαστε σκληρά αλλά με τρόπο δίκαιο νομίζω στις ε, συνεδριάσεις αυτές ε, και στοχευμένα και θα χαιρόμουν. Άρα κύριε Πρόεδρε στο τέλος της σημερινής συζήτησης να δείτε την ε, πρόταση που έχουμε κάνει για να ψηφίσουμε 21 ε, Φεβρουαρίου, να το επισημοποιήσετε για να μπορέσουμε να οργανωθούμε και εσωτερικά στις ε, κοινοβουλευτικές ομάδες για να έχουν όλοι οι βουλευτές την δυνατότητα να δουν τα συμβαστικά κείμενα που υπάρχουν. Ευχαριστώ. Η κυρία Χόλ έχει λοιπόν το λόγο. Thank you. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για το έργο που έχει φέρει σε πέρα στο θέμα αυτό και οι σκιές μου, οι σκιώδες εισηγητές μου δηλαδή, θα συμφωνήσουν ότι έχουμε κάνει πολύ εργασία, εργασία σκαπανέως για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε όλα τα προβλήματα που υπήρχαν στο κείμενο, το οποίο διεξήλθαμε παράγραφο προς παράγραφο. Έχουμε επιτύχει σημαντική πρόοδο, πιστεύω. Γιατί παρά το γεγονός ότι υπήρχαν πολλά ανοιχτά πολιτικά θέματα που φυσικά θα μας χώριζαν σε πολιτικές παρατάξεις. Νομίζω ότι έχουμε αρχίσει να αποδεικνύουμε οι μεν στους δε και τούμπαλιν ότι μπορούμε να έχουμε ένα αποδεκτό επίπεδο συνένεση. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα λοιπόν τον εισηγητή για τη διαδικασία αυτή, την οποία εγώ υποστηρίζω απόλυτα, όπω υποστηρίζω και αυτά τα οποία προέτεινε σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα. Πιστεύω ότι αν συνεχίσουμε το έργο μα όσο έχουμε πράξει μέχρι τώρα με ένα συστηματικό τρόπο, τότε θα μπορέσουμε να δώσουμε την πρέπουσα προσοχή σε όλα τα τμήματα της οδηγίας. <clears throat> Χαιρετίζω επίσης την δήλωση της Κομισιόν που μόλις τώρα έγινε. Με καθησυχάζει οι διαβεβαίωση που δώσανε για τους δημόσιους διαγωνισμούς και τις δημόσιες προμήθειες. <clears throat> Γιατί μας ενδιαφέρει να συμπεριληφθεί και, αυτό το, και αυτή η μνήα στο έγγραφο. Για την τιμολόγηση, εγώ μόλις ήρθα από ένα πρόγευμα εργασίας με θέμα το τι μπορεί να δώσει στους καταναλωτές η ευφύης τιμολόγηση. Ένας από τους τομείς που έχουμε συζητήσει πάρα πολύ ως σκιώδεις εισηγητές και ελπίζω ότι μπορώ να μεταφέρω και την άποψη των συναδέλφων λέγουσα ότι υπάρχει η έντονη εντύπωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι είναι πάρα πολύ σημαντική για τους καταναλωτές αυτή η οδηγία να μπορέσει να ευδοκιμήσει και να λειτουργήσει και θα πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στους εκλογείς μας και θα πρέπει να έχουν πληροφορίες, συμβουλές και να αποκομίσουν τα πλεονεκτήματα της τιμολόγησης από εξατομικευμένους μετρητές. Χαιρετίζω επίσης αυτά που είπε η Κομισιόν για τους στόχους που επιζητεί. Το πιο σημαντικό στις συζητήσεις μας είναι να κρατήσουμε στο προσκήνιο πάντα τους λόγους που μας οδηγούν στο να αντιμετωπίσουμε αυτό το νομοθέτημα και τους λόγους οι οποίοι μας οδηγούν σε ένα στόχο 20% για την ενεργειακή βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, το οποίο σημαίνει και ένα συγκεκριμένο ποσό εξοικονομούμενης ενέργειας. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να ελέγξουμε την κλιματική αλλαγή και να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε και μια καλύτερη παροχή ενέργειας στην Ευρώπη και τους καταναλωτές. Κάποιες ακόμα παρατηρήσεις που θα ήθελα να κάνω. Γενικά, το κείμενο της Κομισιόν ήταν δύσκολο να το αποδεχτούν ορισμένα κράτη-μέλη, γιατί τα κράτη-μέλη τα οποία ήδη είχαν αναλάβει δράση σε πολλούς τομείς ενεργειακής απόδοσης, είδανε ότι αυτά τα οποία προτείνει η Κομισιόν δεν συναρμοζόταν πλήρω με αυτά τα οποία είχαν πράξει ήδη στο παρελθόν. Ίσως λοιπόν θα μπορούσαμε να σκεφτούμε τη δυνατότητα να έχουμε μεγαλύτερη ευελιξία στο κείμενο. Αυτό είναι κάτι το οποίο το εξετάσαμε ω κοιόδη συζητητέ, ώστε ενώ επιζητούμε και επιτυγχάνουμε του ίδιου στόχου και τι ίδιε φιλοδοξίε, σε τελική ανάλυση, θα μπορούσε αυτό να μας δώσει τη δυνατότητα να εκμεταλλευτούμε και τις εθνικές μας πρωτοβουλίες και όχι να ξεκινήσουμε από το μηδέν. Νομίζω ότι έχουμε ήδη πετύχει σημαντική πρόοδο στην επιτεύξη αυτή τη ευελιξία. Τέλο, ένα άλλο τομέα για τον οποίο νομίζω ότι μπορούμε να δώσουμε σωστή έμφαση είναι αυτό ο τομέα που αφορά τι μικρομεσαίες επιχειρήσει. Όλοι κατανοούμε τη σημασία <clears throat> των επιχειρήσεων αυτών μέσα στα πλαίσια της τωρινή οικονομικής συγκυρίας και της κρίσης, κάτι το οποίο προτείνουμε στην οδηγία, είναι και η εξαίρεσή τους από τους ενεργειακούς ισολογισμούς και το να μπορέσουν να τεθούν σε λειτουργία και μέτρα ευνοϊκά για τις εταιρείες αυτές που όχι μόνο θα βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση αλλά θα μειώσουν και το κόστος το οποίο επομίζονται για την εξοικονόμηση ενέργειας νομίζω ότι θα μπορέσουμε με τον τρόπο αυτό να συνεχίσουμε να δίνουμε έμφαση στην πτυχή αυτή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που εξακολουθεί να είναι πάρα πολύ σημαντική σε μια δύσκολη οικονομική κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Έχουμε πολύ δρόμο να διατρέξουμε ακόμα. Για μένα όμως το πιο σημαντικό είναι ότι έχουμε ξεκινήσει αυτό το ενδελεχές έργο εξέταση κάθε παραγράφου και ελπίζω θα μπορέσουμε να το περατώσουμε αυτό το έργο. Ο κύριος Πίπα. <coughs> Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να επενέσω τον εισηγητή για, την, ε, για τον εργόδη τρόπο με τον οποίο έχει αντιμετωπίσει αυτό το νομοθέτημα και για την πολύ καλή εργασία του. Έχουμε συνεργαστεί μαζί του όλοι και πιστεύω ότι έχουμε καταφέρει να βρούμε συμφωνίες σε πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία. Ίσως όχι ακόμα στα αποφασιστικά σημεία βέβαια. Θα ήθελα να τονίσω ότι στο άρθρο 2 που αφορά τα χρηματοδοτικά μέσα βρισκόμαστε σε καλό δρόμο. Το ίδιο ισχύει και για το άρθρο 10 το οποίο θέλει να θέσει πιο πολλά οικονομικά στοιχεία στη συμπαραγωγή ενέργειας και ισχύω. Και επίσης χθες καταφέραμε να πετύχουμε και περισσότερες ε, συμφωνίες για το σημείο 7, δηλαδή τους ενεργειακούς ελεγχούς και ισολογισμούς και επίσης για το σύστημα πιστοποίησης για την ε, αναγνώριση της, ε, της ενεργειακής απόδοσης, τον καθορισμό λοιπόν των συστημάτων αυτών. Και ο στόχος μας φυσικά δεν είναι να αντικαταστήσουμε τα υφιστάμενα συστήματα μέσα στα κράτη-μέλη με ένα νέο ευρωπαϊκό σύστημα. Και είδαμε την κατάσταση ορισμένων κρατών μελών και σε σχέση με αυτά μπορέσαμε να καταλήξουμε σε κάποια συνένεση. Σε ό,τι αφορά τώρα την ε, γνωμοδότηση της Επιτροπής ε, Περιβάλλοντος, θα ήθελα να ξέρω και ποια είναι η άποψη του εισηγητή για τη γνωμοδότηση αυτή. Το ΕΛΚ από τη δική του πλευρά έχει κάνει μια σειρά από αρκετά ευέλικτες ε, προτάσεις τροποποίησης, αλλά συγχρόνως τόνισε και την ανάγκη να συμπεριφθεί το σύστημα εκπομπής, εμπορίας εκπομπών αριών του θερμοκηπίου, το ETS. Και θα ήθελα να την απόψη του εισηγητή. Επίσης για το χρονοδιάγραμμα έχουμε συμφωνήσει σε πολλές ε, λεπτομέρειες, αλλά όχι σε όλα τα κέρια και κομβικά θέματα. Πιστεύω ότι το χρονοδιάγραμμα στο μέλλον θα εξαρτηθεί από το βαθμό στον οποίο θα μπορέσει ο εισηγητής να επιτύχει να υπάρξει συνένεση επί τη βάση των προτάσεών του, ιδίως στα άρθρα 3, 4 καθώς και 6. Μέχρι στιγμή δεν έχουμε καταφέρει να συμφωνήσουμε στα σημεία αυτά και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να φτάσουμε σε μια γρήγορη λύση για τα σημεία αυτά, οπότε θα μπορέσουμε να τηρήσουμε και το προτινόμενο χρονοδιάγραμμα. Αυτό όμως εξαρτάται και από τις προσπάθειες του εισηγητού. Μερσή, ο κύριος Βιδάλ Κουάδρας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω και εγώ να καλωσορίσω τον νέο επικεφαλής μονάδας, τον Τσάρς Μπάιερ. Είχα τη χαρά να δουλέψω μαζί του για χρόνια στον τομέα του συμβιβασμού. Έχουμε ζήσει μαζί περισσότερες ημέρες ε, ε, κατά τις οποίες υποφέραμε παρέμερες δόξας. Ε, ελπίζω ότι εδώ θα γνωρίσουμε περισσότερη δόξα σε αυτή την Επιτροπή από τη βάσανα. Κύριε Πρόεδρε, είναι πολύ καλό που αναβλήθηκε κατά ένα μήνα η ψηφοφορία για αυτό το φάκελο. Χρειαζόμαστε χρόνο για να συζητήσουμε τα θέματα που μπορούμε να προωθήσουμε. Έχουμε συζητήσει μια φορά για τις τροπολογίες, αυτή τη φορά τη συζητάμε για δεύτερη φορά. Έτσι θα μπορέσουμε να είμαστε πιο ακριβείς. Όσον αφορά το δίλημα δεσμευτικού στόχου ή πολλών πολυάριθμων δεσμευτικών μέτρων, κατά την άποψή μου δεν πρέπει να ε, προσπαθούμε να κερδίσουμε μάχες που δεν μπορούμε να κερδίσουμε. Είναι προτιμότερο να υιοθετήσουμε μια ρεαλιστική προσέγγιση. Μέτρα λοιπόν που θα αποφασιστούν από τα κράτη-μέλη στα εθνικά σχέδια απόδοσης με επίτευξη επιμέρους ε, στόχων που θα έχουν οριστεί από κάθε κρατος μέλος ως αποτέλεσμα αυτής της οδηγίας. Αυτή πιστεύω είναι η ρεαλιστική προσέγγιση σε περίπτωση που τα εθνικά σχέδια προγράμματα δεν ε, επιτύχουν, δεν επιτύχουν τους στόχους τους, σε αυτή την περίπτωση τα μέτρα αυτής της οδηγίας θα εφαρμόζονται με τρόπο δεσμευτικό στα κράτη-μέλη. Και η Κομισιόν φυσικά θα πρέπει να ελέγχει κατά πόσο τα προγράμματα τηρούν ή όχι τους στόχους. Ούτως ή άλλως, σε κάποια περίπτωση δεν πρέπει να διπλασιάζουμε τις υποχρεώσεις ε, υποβολής εκθέσεων. Προτείνω λοιπόν οποιοδήποτε αποκλειών μέσο να υπόκειται στην υποχρέωση του άρθρου του σχετικού άρθρου και τα κράτη-μέλη να πρέπει να αποδεικνύουν ότι τα προγραμματά τους επιτυγχάνουν τον εθνικό στόχο. Όσον αφορά το άρθρο 3, επιμένω στο σημείο που ανέφερα την προηγούμενη φορά, να διατηρήσουμε το άρθρο όπως το προτείνει η Κομισιόν, αλλά να λέμε και ξεχωριστά ότι όσον αφορά το μίσ της βιομηχανίας μας με υψηλή κατανάλωση ενέργειας, τα κράτη-μέλη πρέπει να έχουν στόχο όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας ε, από άποψη ΑΕΠ την ένταση ουσιαστικά ενέργειας με την ενέργεια της κατανάλωσης. Το έχω πει πολλές φορές ότι πρέπει να συμπεριλάβουμε όλους τους τρόπους συμπαραγωγής και πρέπει να αναπτύξουμε τη συμπαραγωγή ε, θερμότητας και ηλεκτρισμού όχι υποχρεωτικά αλλά μόνο όταν τεχνολογικά είναι εφικτό αυτού του είδους οι γενικές υποχρεώσεις μπορεί να οδηγήσουν σε αντιπαραγωγικά αποτελέσματα σε ορισμένε περιπτώσεις. Στη σχέση που αναφέρεται στα άρθρα 4 και 5 συμφωνώ με τον εισηγητή ότι εκτός από την ανακαίνιση κτηρίων ε, τα κρατημέλη μπορούν να λάβουν επιπλέον μέτρα που θα μειώνουν την κατανάλωση κάθε χρόνο. Μπορούμε να διαπραγματευτούμε το ποσοστό για αυτά. Ο εισηγητής προτείνει 3%. Εμείς μπορούμε να το συζητήσουμε κατά πόσο θα είναι 3% ή κάποιο άλλο ποσοστό. Ωστόσο, επί της αρχής συμφωνούμε. Η αρχή είναι ότι η ενεργειακή απόδοση των κτηρίων μπορεί να βελτιωθεί μέσω της ανακαίνησης αλλά και μέσω υπηρεσιών ενεργειακής απόδοσης όπως ε, επιμέρους μετρητές και άλλα μέτρα. Για να ολοκληρώσω κύριε Πρόεδρε θα ήθελα να επιμείνω στην αρχή ότι πρέπει πραγματικά να επιμείνουμε στα μέτρα διαχείρισης βάσει της ζήτησης. Επανειλημμένως έχω, επαναλα... έχω τονίσει σε αυτή την Επιτροπή ότι τα μέτρα που επικεντρώνονται στη ζήτηση και οι σχετικές υπηρεσίες και οι συσκευές μέτρησης συμβάλλουν σημαντικά στην ενεργειακή απόδοση όχι μόνο μειώνουν σημαντικά την πίεση προς το grid, προς το δίκτυο, αλλά έχουν και τη δυνατότητα να το επιτυγχάνουν με προσέγγιση επικεντρωμένη στην αγορά, που είναι σε όλες τις περιπτώσεις η καλύτερη προσέγγιση, η προτιμότερη προσέγγιση σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Κύριος Γκίρεκ. Ευχαριστώ πολύ πρώτα απ' όλα ε, θα ήθελα να πω το πόσο συμφωνώ με τον κύριο Βιδάλ Κουάντρας. Είναι πραγματικά απαραίτητο να αφαιθεί στα κράτη-μέλη του πώς θα επιτύχουν τους στόχους αυτής της αποτελεσματικότητας και όσον αφορά το ΑΕΠ αυτό έχει ζωτική σημασία Κυρίε και κύριοι, δεν ισχύει το ότι ο χρόνος ε, πιέζει. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα για να το ξεπετάξουμε. Οπότε όσο πιο πολύ μας απασχολήσει τόσο το καλύτερο. Είχε γίνει μια λανθασμένη αρχή γιατί βεβαίως δεν ξέραμε τι ήταν η ενεργειακή ε, αποδοτικότητα. Είτε για τους τομείς είτε για τις χώρες δεν είχαμε ορισμό. Όταν μιλάμε για τις χώρες πρέπει να είναι ορισμός του ΑΕΠ αυτός ο οποίος ισχύει. Και βεβαίω ο ορισμός πρωτογενούς ενέργειας επίσης δεν ήταν σαφής. Εγώ έχω κάνει τη δική μου έρευνα και βρήκα διάφορους ορισμούς. Κύριε Τούρμες, η ανανεώσιμη ενέργεια είναι πρωτογενής ενέργεια ή όχι και πώς μετράει κανείς την αποτελεσματικότητα. Αυτά μπορεί να ακούγονται λεπτομέρειες, αλλά έχουν ε, ζωτική σημασία. Νομίζω πως η ηλιακή ενέργεια είναι η πρωτογενής ε, πηγή ενέργειας ε, κατεξοχήν. Κάτι ακόμα. Νομίζω πως πρέπει να αναβληθεί αυτό το θέμα, αλλά Πρέπει επίσης να δοθεί δυνατότητα να έχουμε περισσότερες τροπολογίες. Οι 1800 ε, τροπολογίες εδώ πέρα οφείλονται κυρίως σε παρεξήγηση. Δεν υπάρχει σαφήνεια για πολλά πράγματα. Οπότε, εάν είναι δυνατόν ε, από τη δικαστική απόψη, εγώ θα ήθελα να καταθέσουμε και άλλες τροπολογίες. Η κυρία Ντελκαστήγιο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να θα τράξω αυτή την ευκαιρία για να ευχαριστήσω για να ευχηθώ μάλλον καλή χρονιά σε όλους τους παρόντες και θα έρθω στο θέμα. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε ότι βρισκόμαστε σε μια διαδικαστική φάση όπου έχει ήδη εκπνεύσει η προθεσμία για την παρουσίαση τροπολογιών. Επομένως, οποιαδήποτε συμφωνία θα πρέπει να γίνει επί τη βάση των τροπολογιών που έχουν ήδη κατατεθεί. Υπάρχει φυσικά ένα ευρύ περιθώριο ακόμα γιατί υπάρχουν τροπολογίες οι οποίες είναι αρκετά διαφορετικές μεταξύ τους και επομένως η τέχνη της σύναψης συμβιβασμιστικών λύσεων θα εξαρτηθεί πολύ από την ικανότητα του εισηγητή, τον οποίο θέλω να ευχαριστήσω φυσικά και για το έργο που έχει κάνει, τον Κλάβδιο Τόρμες και επίσης και όλους τους σκιώδεις εισηγητές. Υπήρξε επίση και η αφοσίωση πολλών συναδέλφων οι οποίοι παρακολουθούν αυτό το θέμα, ένα θέμα το οποίο ενδιαφέρει πάρα πολλού βουλευτέ και υπάρχει μεγάλη συμμετοχή από τα μέλη αυτή τη επιτροπή, στην εκπόνηση λύσεων συμβιβαστικών και όλα αυτά. Τώρα, δεδομένου ότι υπάρχουν πολλέ δυνατότητε ανοιχτέ μπροστά μα. εγώ θα ήθελα να αναφερθώ μονάχα σε δύο επιλογέ. Η πρώτη επιλογή έχει να κάνει με την ευελιξία των μέτρων που θέλουμε να θεσπίσουμε εδώ. Είναι κεφαλαιόδες, <clears throat> να μπορεί να υπάρχει δυνατότητα επιλογής προαίρεσης από τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν τα μέτρα που θεωρούν πιο πρόσφορα για να πετύχουν τους, τους στόχους τους. <clears throat> σε αντίθετη περίπτωση θα αποτύχει αυτή η διαδικασία, όπως και σε πολλά άλλα νομοθετήματα, τα οποία στη συνέχεια ξενερώνονται για να μπορέσει να αποφύγει ε, ένα κράτος μέλος <clears throat> για να δεσμευτεί από αυτά δεν είναι καλό νομοθέτημα, ένα νομοθέτημα το οποίο δεν εφαρμόζεται σωστά. Και γι' αυτό πρέπει να είμαστε ρεαλιστέ. Η κατάσταση των κρατών μελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ ποικιλή. Γνωρίζοντα λοιπόν αυτό, δεν πρέπει να επιμείνουμε να υπάρξει ένας ενιαίος στενός κορσέ για όλους και να υπάρξει και η ίδια πορεία δράση από όλου. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο είναι καθοριστικό γιατί αυτό το στοιχείο θα προσδιορίσει στο μέλλον το μέλλον αυτής της οδηγίας και την αποτελεσματικότητα εφαρμογής της στον τομέα της ενεργειακής κατανάλωσης. Τούτου λεχθέντος, εγώ θα ήθελα να επιμείνω να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω. Υπάρχουν ορισμένα μέτρα, όπως αυτά τα οποία συνάπτονται με την ανακαίνιση των κτηρίων και την εφαρμογή ενεργειακών μέτρων στα κτίρια αυτά, καθώς και μία πλειάδα μέτρων προσθέτων που εξαρτώνται από τη δράση του δημοσίου τομέα. Κάτι ακόμα όμως πρέπει να σας τονίσω. Στην Ισπανία να γνωρίζετε ότι στα δημόσια κτίρια, τα οποία βέβαια δεν είναι καινούργιες κατασκευές, ή για άλλους λόγους που υποχρεώνει την, ε, τον κάτοχο του κτηρίου να ανακαινήσει το κτίριο αυτό, για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ε, ό,τι και να λέει οδηγία, επειδή θα αλλάξουν πολύ τους γλόμπους, παραδείγματος χάρη, φωτισμού, της, ε, της λιχνίας φωτισμού και θα θέσουν λιγότερο ενεργοβόρες ε, ε, λαμπτήρες και επομένως θα υπάρξει ούτως ή άλλως μια επένδυση προς την κατεύθυνση αυτή, εφόσον υπάρχουν τροπολογίες προς την κατεύθυνση αυτή, θα πρέπει να υπάρξει μια συμφωνία, ώστε όταν μια χώρα δεν μπορεί γιατί πρέπει να καλύψει τους στόχους του ελλείμματός του, επειδή φέρει σε πέρας μια σειρά από μέτρα για δημοσιονομικού χαρακτήρα και επίσης λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι πρέπει να υπάρξει και συμμόρφωση με τον εθνικό προϋπολογισμό και τις επιταγές της Κομισιόν. Όταν λοιπόν τα κράτη-μέλη μπορούν να προβάλλουν ότι υπάρχουν λόγοι δυσκολίας εφαρμογής αυτής της οδηγίας για λόγους προϋπολογισμού ή για άλλους λόγους. <clears throat> Γιατί είναι πολύ πιο σημαντικό να καλύψουμε στόχους υγειονομική περίθαλψη ή παιδεία παρά να εφαρμόσουμε στόχου ενεργειακή απόδοση, τότε θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα κάποια εξαίρεση. Αυτό είναι ένα στοιχείο τη πραγματικότητα. Αν δεν το κατανοήσουμε αυτό και αν δεν κατανοήσουμε τη γενική ανάγκη ευελιξία όλων αυτών των μέτρων, είμαστε πολύ μακριά από την μπάλα, είμαστε πολύ μακριά από την πραγματικότητα. Το να μιλήσω εγώ τώρα στου Ισπανού και να πω ότι πρέπει να γίνουν <clears throat> όλα αυτά τα πράγματα που προβλέπει αυτό το νομοθέτημα, αυτό του δίνει την εντύπωση ότι εγώ ω κοινοβουλευτικό και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο οποίο συμμετέχω ότι είναι σε άλλο πλανήτη. Και σας το λέω αυτό ότι <clears throat> πρέπει να το κατανοήσετε αυτό γιατί είμαστε υποχρεωμένοι να αντιμετωπίσουμε την πραγματικότητα πάρα πολλών χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πιστεύω ότι οι εισηγητή και οι σκιωδησίτε έχουν ένα πολύ δύσκολο καθήκον. 1812 τροπολογίε είναι πάρα, πάρα πολλέ. Ίσως θα μπορούσαμε να του βοηθήσουμε. Όπω είπε ο κ. Γκιαρέκ, θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα βήμα πίσω και αυτή επίση και να εξετάσουμε την κατάσταση αυτή από έξω, να ξεκαθαρίσουμε του ορισμού. Πιστεύω ότι πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τις ε, βασικές αρχές σε αυτή την πρόταση. Αυτή είναι η δική μου ιδέα, η δική μου άποψη. Θα ήθελα επίσης να μιλήσω για μια-δυο τροπολογίες. Οι βασικές αρχές ε, ε, που θα ήθελα να αναφέρω. Πρώτον, χρειαζόμαστε ρεαλιστικούς στόχους που είναι εφικτοί. Μπορούμε να είμαστε φιλόδοξοι βεβαίως, αλλά αν ορίσουμε με ρεαλιστικούς στόχους, κανείς δεν θα μας πάρει στα σοβαρά. Και τότε θέτουμε σε κινδύνο και άλλους στόχου τη πρότασης. Η δεύτερη βασική αρχή είναι ότι χρειαζόμαστε ευνοϊκές συνθήκες. Διότι έτσι θα λυθούν πολλά προβλήματα. Ε, υπερβολικά πολύ διοικητικό φόρτος ε, θα είναι επιζημίω και για αυτό και για άλλου τομεί. Θα χρειαστεί λοιπόν να εμπιστευτούμε τη λειτουργία της αγοράς. Η τρίτη βασική αρχή είναι η εξή. Πρέπει σε όλες τις περιπτώσεις να μην ξεχνάμε ότι τα κράτη-μέλη έχουν αναπτυχθεί σε διαφορετικά επίπεδα. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ. Αυτό μοιάζει με τις δύο πρώτες αρχές. Πρέπει πάντα να έχουμε υπόψη μας την πραγματική κατάσταση, να είμαστε ρεαλιστές. Διαφορετικά, μη ρεαλιστικοί κανόνες δεν θα μας οδηγήσουν σε καμία λύση. Αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να αναφερθώ σε τέσσερα ζητήματα που ανέφεραν και κάποιοι άλλοι συνάδελφοι. Το πρώτο είναι η στόχη εξοικονομής ενέργειας. Είμαι πεπισμένος ότι εφόσον ακολουθήσουμε αυτές τις βασικές αρχές θα υπάρχουν διαφορές στην κατανάλωση ενέργειας μεταξύ κρατών μελών. Αν λάβουμε υπόψη όλες αυτές τις διαφορές, σε κάποια κρατημέλη υπάρχουν, υπάρχει ψηλότερη κατανάλωση και υπάρχουν ίσως και άλλες πηγές κατανάλωσης εκτός από τις κατοικίες. Θα χρειαζόμαστε στοχευμένες τιμές λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις διαφορές μεταξύ κρατών μελών. Το δεύτερο, οι έξυπνοι μετρητές. Πιστεύω δεν είναι ρεαλιστικός αυτός ο στόχος το να φτιάξουμε, ε, ε, να εγκαταστήσουμε τέτοιους μετρητές σε κάθε σπίτι και στις 27 χώρες. Πιστεύω ότι οικονομικά δεν είναι βιώσιμο αυτό. Ε, εμποδίζει την επιτευξή του αρχικού στόχου. Χρειάζεται να διεξάγουμε μια ανάλυση κόστους και ωφέλους και να προχωρήσουμε σε αυτό το βήμα όταν θα είναι οικονομικά ωφέλιμο και αποδοτικό. Το τρίτο, η συμπαραγωγή και θέρμανσης και ηλεκτρισμού. Οι κανόνες πιστεύω είναι πολύ περιοριστικοί, παρεμβαίνουν στους μηχανισμούς της αγοράς. Πιστεύω ότι και εδώ πρέπει να χρησιμοποιήσουμε έναν μηχανισμό ε, κόστους και ωφέλους και εφόσον το αποτέλεσμα είναι θετικό από την ανάλυση, είμαι σίγουρος ότι οι παράγοντε τη αγοράς θα λάβουν δράση, θα κάνουν όλα τα βήματα που τους προτείνουμε εφόσον η αγορά αντιδράσει από μόνη της μπορούμε να, το αφήσουμε, να την αφήσουμε να κάνει ό,τι θέλει και να αποφύγουμε να δημιουργήσουμε μια προγραμματισμένη οικονομία διότι κοιτώντα τα παραρτήματα αυτή τη στιγμή αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και το τέταρτο που ήθελα να πω είναι το, ο στόχος του 3% για την ανακαίνιση των δημοσίων Πρέπει να γνωρίζετε ότι αυτή τη στιγμή ο στόχος ανακαίνισης είναι κάτω από το 0,5% ε, στα περισσότερα κράτη-μέλη. Να, το να περάσουμε από το 0,5% στο 3% ουσιαστικά είναι μη ρεαλιστικό. Ακόμη περισσότερο αν ε, αναλογιστούμε την τρέχουσα οικονομική ε, κρίση. Είναι εξαιρετικά δύσκολο αυτό που πρέπει να σκεφτούμε. Είναι το πώς θα δημιουργήσουμε ευελιξία για τα κράτη-μέλη και πώς μπορούμε να τα βοηθήσουμε να δημιουργήσουν τη δική του συμβουλή. Έχω μια συγκεκριμένη πρόταση με στόχο την έβρεση ε, συμβιβασμού στην Επιτροπή μας και μετά στο Συμβούλιο. Όσον αφορά αυτή τη συμβολή των ιδιοκτητών, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το πλεόνασμα των ποσοστώσεων και να χρησιμοποιήσουμε αυτό τα έσοδα για να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη να το χρησιμοποιήσουν ως δική του συμβολή. Αυτό μας φέρνει πιο κοντά στο συμβιβασμό. Για να κλείσω, επιτρέψτε μου να πω κύριε Πρόεδρε, ότι πρέπει να είμαστε ρεαλιστικοί και να εμπιστευτούμε τις αγορές. Αυτή θα είναι η, η η βασική οδός που θα μας οδηγήσει σε κάποια λύση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Έχω 8 ακόμα που πρέπει να λάβουν το λόγο. Συγγνώμη που σα ε, δείχνω την αδειμονία μου και είναι και η Κομισιόν πρέπει να λάβει το λόγο. Σα παρακαλώ λοιπόν να συντομεύετε λιγάκι αυτά τα οποία θέλετε να πείτε. Καταλαβαίνω ότι είναι σημαντικό αυτό το, πολιτικό, το θέμα αυτό από πολιτική άποψη. Η κυρία Νίμπλα. Ωραία. Ό,τι πείτε κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα καλή χρονιά και από μένα. Και βεβαίως ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή μας, τον Κλοντ μας και όλους τους κοιόδης εισηγητές. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό το πόσο γρήγορα βρίσκουμε συμβασμούς για 1800 ε, τροπολογίες και πραγματικά αξίζει σεβασμό ο συνάδελφος. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δουλειά σας. Τρία θέματα θα ήθελα να αναφέρω, μια που έχει προχωρήσει ο χρόνος. Πρώτα απ' όλα η συζήτηση για το θέμα δεσμευτική στόχη, δεσμευτικά μέτρα. Δεν θα σας προξενήσει έκπληξη το ότι όπως και άλλοι συνάδελφοι από τη δική μου και άλλες ομάδες θα πρέπει να υπάρχει, μη, θεωρούν πως θα πρέπει να υπάρχει απαραίτητη ευελιξία για να μπορέσουμε να πούμε ναι εντάξει δεσμευτική στόχη αλλά όχι δεσμευτικά μέτρα. Ειδικά όταν μιλάμε για υποχρεώσεις στον ε, δημόσιο τομέα, νομίζω πως ε, δεν υπάρχει ανοχή ούτε στους ενδιαφερομένους ούτε στον λαό γενικά και νομίζω αυτά τα οποία πρότεινε ο κύριος Βιδάλ Κουάδρας είναι ένας, ε, μια, ένας εξαιρετικός συμβιβασμός, δηλαδή να ορίσουμε τους στόχους και αν αποτύχουν αυτοί να κάνουμε τα μέτρα δεσμευτικά. Δεύτερη παρατηρήση. Είδα τον συμβιβασμό για το άρθρο 4 και εκεί πέρα διαπίστωσα πρώτα απ' όλα πως ολόκληρο το άρθρο 4 στη νέα του αυτή εκδοχή ε, θέλει να επεκτείνει την υποχρέωση του δημοσίου τομέα και στα κτίρια που νοικιάζει και όχι μόνο κατέχει ο δημόσιος τομέας Occupied by Bagel Bodies, δηλαδή τα κτίρια που νοικιάζει ο δημόσιος τομέας. Αυτό είναι τρέλα. Και δε, δε, πώς θα γίνει αυτό στην πράξη. Δεν μπορούμε να υποχρεώσουμε τον ενοικιαστή να εφαρμόσει υποχρεώσεις ε, του ιδιοκτήτη τελικά ενός κτηρίου. Ούτε λογικό δεν το βρίσκω, ούτε να μπορεί να γίνει. Γιατί σε τι θα οδηγήσει αυτό. Είτε δεν θα νοικιάζει πλέον ο δημόσιος τομέας γιατί θα έχει υποχρεώσεις ιδιοκτήτη ή θα ανέβει τόσο πολύ το νίκη ε, λόγω αυτών των υποχρεώσεων. Ε, θέλω να δω δηλαδή πώς, πώς το φαντάζεστε να γίνει στην πράξη. Εγώ δεν το βρίσκω καλή ιδέα. Τελευταίο σημείο με ικανοποίησε στο συμβαστικό κείμενο του άρθρου 4 παράγραφος 3α αυτό το οποίο γράφει εδώ πέρα. Για να δω ακριβώς τη διατύπωση. Αντί να πάμε σε υποχρεωτική ανακαίνιση, να έχει την δυνατότητα να εξοικονομήσει ένα ποσοστό της χρήσης ενέργειας. Αυτό ακριβώς είναι η ευελιξία που χρειαζόμαστε για να φτάσουμε στον επιθυμητό στόχο. Νομίζω αυτό είναι το σωστό, είναι θαυμάσια ιδέα και θέλω να το στήριξω. Και βεβαίως ε, για το ποσοστό τώρα αν θα πάει πάνω ή κάτω, εντάξει μπορούμε να το συζητήσουμε. Να ευχαριστήσω λοιπόν όλους οι συναδέλφους εδώ και εβδομάδες ασχολούνται εντατικά με αυτό τον φάκελο, τους συμβαστικές προτάσεις και αναμένω τη συζήτηση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Να πω κάτι έτσι ως παράκληση στις συμβαστικές ε, τροπολογίες. Υπάρχουν βουλευτές εδώ πέρα που θέλουν πολύ αυστηρίους ε, κανόνες, κάποιοι συνάδελφοι θέλουν πιο ευέλικτους κανόνες. Συμβιβασμός ε, δεν μπορεί να είναι το αυστηρό να γίνει αυστηρότερο, έτσι ως υπόμνηση, αν θέλετε. Νόρμπερτ Λάγκε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, θα είμαι σύντομος, συμφωνώ με τους ε, συναδέλφους που προλάλησαν. Ε, χαίρομαι εντωμεταξύ για το ότι έγιναν πιο σαφή τα πράγματα όταν μιλάμε για ενεργειακή αποτελεσματικότητα. Ε, ενεργειακή αποτελεσματικότητα σημαίνει και εξοικονόμηση ενέργειας. Εντάξει, βλέπετε, έχουμε μία ύφεση και αυτομάτως υπάρχει εξοικονόμηση ενέργειας σε καιρούς λοιπόν ε, οικονομικών δυσκολιών ε, των κρατών μελών μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την ευελιξία, να χρησιμοποιηθούν τα μέτρα εκείνα τα οποία είναι πιο οικονομικά. Τέλος πάντων τώρα δεν ε, είναι η ώρα για μια συζήτηση αρχών. Δεσμευτικοί στόχοι είναι χρήσιμοι, δεσμευτικά μέτρα μπορούν να είναι αντιπαραγωγικά. Και Ξέρετε, συμβασμό σημαίνει να υποχωρήσουν λίγο και οι δύο για να μπορέσουν να συναντηθούν ε, κάπου στη μέση. Θα πρέπει λοιπόν να το συζητήσουμε για να μπορέσουμε όντω να ε, ψηφίσουμε τον Φεβρουάριο. Θεωρώ πως ε, οι διαφορές που υπάρχουν στα κράτη-μέλη και στα κτίρια μέχρι στιγμής όσον αφορά και την κοινή, τη συνδυασμένη θέρμανση το ανέφερε και ο κύριος Βιδαλκουάδρας, είναι μεγάλες. Ε, τόσο απασχολεί αυτό το ζήτημα και το Συμβούλιο αυτή τη στιγμή. Και αυτή τη στιγμή οι θέσεις απέχουν αρκετά από αυτά τα οποία προτείνει η Δανέζικη Πρόεδρε. Και εγώ είμαι φιλόδοξος, αλλά τόσο αισιόδοξο δεν είμαι. Αυτά και ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Τόμψεν. Ε, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Έχουμε ζητήσει τώρα τα θέματα της ενεργειακής εξοικονόμησης, την ε, εκπροσώπηση των καταναλωτών, των βιομηχανικών κύκλων. Στις, ε, έχουμε ακούσει από απόψεις όλων των εμπειρογνωμών και έχουμε κάνει πολλές συναντήσεις των σκιωδών εισηγητών. Νομίζω ότι κάθε μέρα πλησιάζουμε όλο και περισσότερο σε μια καλύτερη λύση. Παραμένω ακόμα ορισμένα εμπόδια τα οποία πρέπει να ξεπουραστούν, αλλά είμαι πάρα πολύ θετική ότι μπορούμε να φτάσουμε στο στόχο της ψηφοφορία στην Επιτροπή μας το Φεβρουάριο. Αυτό μας δίνει επαρκή χρόνο για να επιτύχουμε μια ευρεία συνένεση και καλά αποτελέσματα που να είμαστε υπερήφανοι για αυτά τα αποτελέσματα. Τι είναι αυτό που δεν καταλαβαίνουμε σε αυτή τη συζήτηση εδώ. Είναι οι λέξεις ρεαλιστική στόχη. Έχουμε στόχους. Οι στόχοι όμως δεν αντικείμενο συζήτηση αποφασιστήκαν στις 12 Δεκεμβρίου από το Συμβούλιο και μετά από το Κοινοβούλιο το 2008 λέω, όχι το 2011 μέσα στα πλαίσια των στόχων του 20-20-20 για το 2020. Το 20% αύξησης της ενεργειακής απόδοσης ήταν δεσμευτικός στόχος. Γιατί είπαν τα κράτη-μέλη μπορούμε να το πετύχουμε χωρίς δεσμευτικούς στόχους, αλλά δεν έχουν πετύχει τίποτα. Ο στόχο όμως υπάρχει. Γιατί μιλάμε τότε για ρεαλιστικού στόχους. Στην Ευρώπη έχουμε ευρωσκεπτικισμό. Γιατί. Γιατί παίρνουμε αποφάσεις οι οποίες δεν εκπληρούνται, δεν εφαρμόζονται στην πράξη. Μη με ρωτήσετε πότε θα αρχίσετε να εφαρμόζετε αυτά τα οποία αποφασίσατε το 2008. Και τώρα λέμε για ρεαλιστικού στόχους. Μα έχουμε στόχους. Αυτό το οποίο συζητάμε σε αυτή την οδηγία και αυτό για το οποίο πρέπει να βαστάσουμε σε μια συμβαστική λύση είναι πώς θα πετύχουμε τους στόχους, όχι αν είναι ρεαλιστικοί. Με ένα πιο εύκαμπτο τρόπο, με κάποιο διαφορετικό τρόπο για κάθε κάτω μέλο, αλλά ο στόχος είναι εκεί πέρα. Το να ξεκινήσουμε μια συζήτηση για ρεαλιστικούς στόχους, όχι, έχουμε δεσμευτεί για μία εξοικονόμηση 20% μέχρι το 2020. Πιστεύω ότι για να πετύχουμε το στόχο χρειαζόμαστε να έχουμε δεσμευτικά μέτρα, δεσμευτικούς στόχους και υπήρξε μια πλειοψηφία στην Επιτροπή μας για τη θέσπιση υποχρεωτικών στόχων. Δεν μπορούμε να χωρίσουμε λοιπόν, να διαχωρίσουμε τους δεσμευτικούς στόχους και τα δεσμευτικά μέτρα, γιατί τα μεν συμπληρώνουν τους δε. Είναι σημαντικό επίσης να έχουμε και κάποιο περιθώριο παραχωρήσεων στον τριγωνικό διάλογο. Μα είπε και η Κομισιόν ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα, διότι είναι διαφορετική στάση στο Συμβούλιο από τη στάση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θέλουμε λοιπόν δεσμευτικού στόχου και υποχρεωτικά μέτρα για να υποστηρίξουν του στόχου αυτού. Για το ερώτημα του αν αυτή η οδηγία θα πρέπει να θέσει όχι μόνο στόχου αποδοτικότητας αλλά και κατανάλωση και ένταση ενέργεια. για μένα δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι για να φτάσουμε το στόχο της αποδοτικότητας θα πρέπει να έχουμε και στόχους μείωσης της κατανάλωσης και αυτό συμπεριλαμβάνει και την χρησιμοποίηση της συμπαραγωγής σε μεγαλύτερο επίπεδο στα άρθρα 11 και 12. Η κατανάλωση αυτή καθεαυτή έχει να κάνει μονάχα με την ε, οικονομική συγκυρία. Και αν βασιζόμαστε μονάχα στην κατανάλωση δεν θα κάνουμε πιστευτό το να επιτύχουμε το στόχο της μείωσης 20%. Έχουμε διαπραγματευτεί Συμβαστικέ τροπολογίε στα άρθρα 7, 8, 9 και 10 και πλησιάσουμε τώρα σε μια συμφωνία η συμβαστική λύση για το άρθρο 8 είναι αυτή η οποία με γεμίζει με περισσότερη ευτυχία. Για, τα, για τους ευφυείς μετρητές. Υπάρχουν πολλές συζητήσεις για τους μετρητές αυτούς στην Ευρώπη. Αλλά εξέφρασε τη θέση του το Κοινοβούλιο όταν ψηφίσαμε για το τρίτο πακέτο για την εσωτερική αγορά ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είπαμε το 2019 πρέπει να έχουν εφαρμοστεί οι εφείς αυτοί μετρητές στην Ευρώπη. Και υπάρχει τώρα μια συμβαστική τροπολογία για το άρθρο 8 που εξασφαλίζει ότι όσο δεν μπορούν οι καταναλωτές να αντιδρούν σε μία αλλαγή των τιμών τιμολογίων ενεργείας σε πραγματικό χρόνο θα πρέπει να παρεμβαίνει και η Κομισιόν. Και είπαμε ότι όταν χρησιμοποιηθούν και αυτοί οι ευφυείς μετρητές θα υπάρχει και προστασία των καταναλωτών και των δεδομένων ώστε μόνο οι καταναλωτές να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα όποτε το επιθυμούν. Υπάρχουν πολλά ακόμα μπορούμε να πούμε για τις τροπολογίες αλλά θα προτιμήσω να τα συζητήσω λεπτομερώς με τους άλλου χειώδεις εισηγητέ. Για να πετύχουμε όμω μια συμβαστική λύση, είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε για το τι μιλάμε. Κύριε Κύρεκ, <clears throat> όταν είπατε ότι συμφωνείτε με τον Αλέκο Βινταλ λέει ο κύριο Βινταλ <clears throat> ότι θέλει να εστιάσει στην πλευρά της συζήτηση, ενώ εσείς μιλάτε περισσότερο για την πλευρά της προσφοράς, την πλευρά της παραγωγής. Δεν είναι λοιπόν σαφή τα πράγματα. Ευχαριστώ. Έχω όλο και πιο μεγαλύτερο πρόβλημα. Ακόμα περισσότεροι θέλουν να λάβουν το λόγο τώρα. Παρακαλώ. Να κλείσω τον κατάλογο των αγοριτών Αυτή είναι η πρώτη μου πρόταση. Δεύτερον, να προσπαθήσουμε να περιοριστούμε σε ένα με δύο λεπτά ο καθένας και βλέπω τώρα τον κύριο Τόιρερ, ο οποίος έχει γενέθλια και τον συγχαίρω. Ο κύριος Τούρμες για διαδικαστικό θέμα. Μέχρι πότε έχουμε χρόνο για τη συζήτηση αυτή. Μέχρι τις 12.30 λέει ο πρόεδρος. Μα είπα στην αρχή, δεν ήταν όλοι παρόντες, ότι προβλεπόταν η συζήτηση αυτή να γίνει μέσα σε μία ώρα. Έχουμε και άλλα σημεία στην ημερήσια διάταξη. Πρέπει να είμαστε και δίκαιοι προς τους άλλους, να δώσουμε και στα άλλα σημεία της ημερήσιας διάταξης χρόνο συζήτησης. Σας παρακαλώ λοιπόν να παραμείνετε στα 15, στα, στο 1,5 λεπτό καθένα, ώστε σε ένα τέταρτο να προσπαθήσουμε να κλείσουμε. Ξέρω ότι είναι σημαντικό το θέμα αυτό, σας παρακαλώ σε αυτό συγκράτηση. Η κυρία Τσίκαου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Γραμματεία και τους συναδέλφους για όλο τους το έργο. Η ενεργειακή αποδόση αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την επίτευξη χαμηλών τιμών για τους καταναλωτές και την καταπολέμηση της φτώχειας. Επίσης, η ενεργειακή απόδοση προσφέρει θέσεις εργασίας και ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη. Έχω υποβάλει μια τροπολογία με την οποία αυτό που προσπαθώ να πετύχω είναι όχι μόνο τα κράτη-μέλη και οι δημόσιες αρχές ε, και τα νοικοκυριά να πρέπει να βελτιώσουν την ενεργειακή τους υπόδοση αλλά να πρέπει να τη βελτιώσουν και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, οι ευρωπαϊκές υπηρεσίες, οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί. Πρέπει να δίνουμε το παράδειγμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πιστεύω ότι όλα τα κτίρια, όλα τα θεσμικά όργανα, όλες οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να ηγούνται στο μέτωπο της ενεργειακής αποδόσης. Επίσης πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη την τεχνική σκοπιμότητα και τη σχέση αποδόσης και κόστους δεδομένων των διαφορετικών κλιματολογικών συνθήκων σε κάθε κράτος μέλος. Επίσης έχω υποβάλει μια τροπολογία όπου ζητώ ευθυγράμμιση των διατάξεων με προηγούμενες οδηγίες όπως την ενεργειακή απόδοση κτηρίων επειδή το τελευταίο που θα θέλαμε θα είναι δύο διαφορετικές οδηγίες με δύο διαφορετικούς ορισμούς για το ίδιο πράγμα. Θα πρέπει να φροντίσουμε να υπάρχει συνοχή στην νομοθεσία μας. Ένα άλλο σημαντικό σημείο κατά την άποψή μου και εδώ συμφωνώ με την κυρία Νίμπλε σαφώς οι δημόσιες αρχές που είναι ιδιοκτήτες κτηρίων, που είναι ιδιοκτήτες κτηρίων. Δηλαδή μιλάμε εδώ για κτίρια τα οποία ανήκουν στις ε, δημόσιες αρχές. Επίσης θέλω να τονίσω τη σπουδαιότητα της χρηματοδότησης της ενεργειακής απόδεσης. Εάν δεν καταφέρουμε να συντονίσουμε, εάν δημιουργήσουμε αντίφαση μεταξύ αυτής της οδηγίας και των κανονισμών για τα διορθωτικά ταμεία και των υπολείπων κανονισμών που προωθούν την ενεργειακή απόδοση, τότε φοβάμαι ότι αυτή η νομοθεσία δεν θα αξίζει ούτε το χαρτί πάνω στο οποίο γράφτηκε. Διότι τα κρατη και οι απλοί άνθρωποι δεν έχουν τόνους χρημάτων για να σπαταλούν στην ενεργειακή απόδοση. Ζητώ λοιπόν από όλους τους συναδέλφους να με υποστηρίξουν σε αυτό το θέμα. Όταν μιλάμε για τα διάφορα ταμεία, για τους διάφορους κανονισμούς, για τα διαρθρωτικά ταμεία και όλα τα υπόλοιπα ταμεία, θα πρέπει επίση να μην ξεχνάμε και αυτόν τον στόχο ενεργειακή απόδοσης. Κλείνω κύριε Πρόεδρε ε, λέγοντας ε, δύο λόγια σε σχέση με την ευφυή μέτρηση. Στη... Ε, έχει περάσει 1,5 λεπτό, είπε ο Πρόεδρος. Πολύ ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, ε, ε, έλεγα ότι πριν από, λίγα, χρόνια στην Ρουμανία ε, οι μετρητές ε, ε σε κάθε διαμέρισμα. Αυτό μόλις έγινε. Και δεν είναι σωστό τώρα να επιβληθούν νέες υποχρεώσεις στους καταναλωτές. Ριέρα Μαδουρέλ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλή χρονιά. Βλέπω ότι ο κύριος Κλάους Βάιερ είναι πλέον μέλος της Γραμματείας της Επιτροπής μας. Θέλω να τον χαιρετήσω και θέλω επίσης να ευχαριστήσω και τον εισηγητή και όλους τους σκιώδεις εισηγητές για την πολύ καλή εργασία που φέρνουν σε πέρας. Θα ήθελα να κάνω τώρα ένα σχόλιο για το άρθρο 10. Είναι προφανές ότι όπως έχει ε, πει και ο εισηγητής και η Κομισιόν, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όσο δυνατόν πιο υποφελώς την ε, θερμότητα που παράγεται από τη συμπαραγωγή. Αυτό είναι δεδομένο. Αλλά παρά τούτο, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι η θερμική σταθμή, ιδίως η σταθμή συμπαραγωγής, θα πρέπει να παίξουν για κάποιο ρόλο υποστήριξης στις ανανεώσιμες ενέργειες, όπως είναι παραδείγματος χάρη η αιωλική ενέργεια. Για να μπορέσει να λειτουργήσει κάτι τέτοιο, αυτή η σταθμή θα πρέπει να προσαρμόσουν την παραγωγή ηλεκτρισμού στις ανάγκες με μεγάλη ταχύτητα και με μια περιοδικότητα βάση των εχμών στην, στις ανάγκες κατανάλωσης ηλεκτρισμού. Μέσα σε αυτές λοιπόν τις συνθήκες, και αυτό είναι απόλυτα ευκταίο, πιστεύω πρέπει να το υποστηρίξουμε, αναρωτιέμαι πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε την παροχή θερμότητος, θέρμανσης σε μια οικιστική περιοχή. Και αυτό πρέπει να το αντιμετωπίσει και η έκθεση. Αν θέλουμε να πετύχουμε το στόχο 20% ανανεώσιμες ενέργειες, ιδίω σε περιοχές που είναι απομονωμένες όπως είναι η Βυρική Χερσόνησος, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να άρουμε όλα τα προσκόμματα για την ε, πρόοδο προς την κατεύθυνση αυτή. Γι' αυτό πιστεύω ότι η τροπολογία συμβιβασμού για το άρθρο 10 θα έπρεπε να συμπεριλάβει και τη δυνατότητα να υπάρχουν εξαιρέσεις τόσο για τους νέους σταθμούς παραγωγής ενέργειας όσο και αυτούς που είναι ανακαινεσμένοι και που έχουν να κάνουν με την υποστήριξη της παροχής ενέργειας η οποία είναι ευμετάβλητη από πηγές ανανεώσιμες όπως είναι η ολική ενέργεια. Ευχαριστώ. Κύριος Κέλλης. Εδώ μιλάμε για την ενεργειακή απόδοση και την εξοικονόμηση ενέργεια και λέμε ότι δεν μπορούμε να έχουμε κάποιους στόχους λόγω της ύφεσης. Σίγουρα το αντίθετο της εξοικονόμησης είναι η σπατάλη και εφόσον εξοικονομεί κάποιος εξοικονομεί. Τέλος, η όλη συζήτηση λοιπόν είναι μια ε, συζήτηση η οποία είναι επικερδής για όλους και όσο το συντομότερο γίνει τόσο το καλύτερο. Ένα κομμάτι της ενέργειας ε, στην Ευρώπη ε, σπαταλάται σε κτίρια και ένα μεγάλο ποσοστό στο φωτισμό. Δεν μπορούμε δηλαδή να έχουμε ενεργειακή απόδοση εκεί, να κάνουμε εξοικονόμηση χωρίς να μας κοστίσει τίποτα. Μην υπερβάλλουμε με την ύφαση. Η υπερθέρμανση του πλανήτη δεν θα σταματήσει λόγω της ύφασης. Ε, οι παγιοί δεν θα σταματήσουν να λιώνουν λόγω της ύφασης. Και εδώ όπου αυτό το ζήτημα απασχολεί τους καταναλωτές και τα κράτη-μέλη, απόδοση σημαίνει εξοικονόμηση, έχει νόημα οικονομικό οι δεσμευτικοί στόχοι είναι καλοί και οικονομικά και καλοί για το περιβάλλον. Μαρινέσκου. Συνάδελφος Μαρινέσκου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει θέσει ένα στόχο και μπορούμε να τον επιτύχουμε με διάφορους τρόπους. Η παρουσία οδηγία επιδιώκει την επιδεύξη του στόχου μέσω της ενεργειακής απόδοσης. Η ένταση της ενέργειας θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως ε, ε, ορόσημο το ότι βελτιώνουμε την ενεργειακή κατάσταση δεν σημαίνει ότι βελτιώνουμε την ενεργειακή απόδοση. Η αύξηση των τιμών του πετρελαίου θα αυξήσει την ένταση της ενέργειας, αλλά όχι την ενεργειακή απόδοση. Ωστόσο, η ένταση της ενέργειας ε, επηρεάζεται επίσης και από τις καιρικές συνθήκες. Ε, ένα αγρόκτημα, για παράδειγμα, και αυτό δεν επηρεάζει την ενεργειακή απόδοση. Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ένα συνδυασμό προϊόντων, ένα, μια μέθοδο με την οποία θα συνδέονται αυτά που παράγουμε με την ποσότητα ενέργειας που καταναλώνουμε. Πιστεύω ότι η στόχη θα πρέπει να είναι δεσμευτική αλλά ότι τα μέτρα θα πρέπει να είναι ευέλικτα. Ευχαριστώ. Κυρία Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πάρα πολύ εν συντομία. Να σας υπενθυμίσω ότι είναι απαραίτητο να δημιουργήσουμε ένα κοινοτικό πλαίσιο για όλα αυτά, αλλά πρέπει να είναι και ευέλικτο, θα πρέπει να σέβεται την αρχή της επικουρικότητας, της αναλογικότητας. Είναι προφανές για μένα ότι τα μέτρα τα οποία προβλέπουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να μείνουν αρκετά ανοιχτά και ευέλικτα στην εφαρμογή τους, ώστε να προσαρμοστούν στις ιδιαιτερότητες του κάθε κράτους μέλους. Να αφήσουμε λοιπόν και περιθώριο για τις εθνικές πρωτοβουλίες και τοπικές πρωτοβουλίες. Οι εθνικοί στόχοι λοιπόν, αν είναι υπερβολικά ε, περιοριστικοί, θα θέσουν προβλήματα σε μια σειρά από κράτη-μέλη. Πρέπει να εξασφαλίσουμε λοιπόν την ευελιξία εφαρμογής όλων αυτών των μέτρων. Έχω καταθέσει μια σειρά τροπολογιών. Θα πρέπει να κάνουμε καλή διάκριση μεταξύ ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας. Επίσης, για να επιτύχουμε το συνολικό αυτό στόχο τον οποίο έχουμε θέσει μου φαίνεται πάρα πολύ σημαντικό, σεβόμενη την επικουρικότητα, να ενισχύσουμε και τους εθνικούς στόχους με την εισαγωγή μιας σαφούς κατανομής άχθους με μεθόδους μέτρησης και επαλήθευσης, την ίδια της Κομισιόν πάντα, και όλα αυτά τα έχω θέσει υπό μορφή τροπολογιών στο άρθρο 3. Πιστεύω εξάλλου ότι είναι σημαντικό να δημιουργήσουμε μηχανισμούς υποχρεωτικούς που βασίζονται στο βαθμό του δυνατού στις, στους στόχους που έχουμε πετύχει για την ενεργεια κατανάλωση κατά μονάδα δραστηριότητας. Για τη συμπαραγωγή επίσης υπάρχουν κάποιες ρήτρες οι οποίες μπορεί να είναι υπερβολικά περιοριστικές μέσα στην πρόταση της Κομισιόν και στον τομέα αυτό μου φαίνεται σημαντικό να αφήσουμε στα κάτι μελη τη δυνατότητα να προβούν σε μια γενικότερη αξιολόγηση των ε, λύσεων που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν για την ε, εξοικονόμηση ενέργειας επί τη βάση μιας ανάλυσης κόστους-οφέλους χωρίς προκαταλήψεις. <clears throat> Και επίσης δεν μου φαίνεται ιδιαίτερα θετικό το να περιορίσουμε τη χρήση χρηματοδοτικών εργαλείων όπως είναι τα συμβόλαια ενεργειακής απόδοσης. Πιστεύω ότι αυτό αντίθετα που χρειαζόμαστε είναι μέγιστη δυνατή ευελιξία σε ό,τι αφορά την επιλογή των μεθόδων που θα προκριθούν για την επιτεύξη της ενεργειακής εξοικονόμησης. Ευχαριστώ. Η κυρία Μέρφης. Μέρκης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συγχαρητήρια στον εισηγητή και τους και εισηγητές για τη δουλειά που έκαναν και σας ευχαριστώ για την προσοχή που δείξατε στην μικροπαραγωγή ενέργειας γιατί έχει μεγάλη σημασία για το μελλοντικό ενεργειακό μας μείγμα. Κατόπιν έχω ένα ερώτημα γιατί μέχρι στιγμής δεν έχω δει συμβαστικές τροπολογίες ε, όσον αφορά τους ορισμούς αλλά μπορεί να μου ξέφυγε κάτι. Θα ήθελα να γνωρίζω τι συνέβη με την ε, επέκταση εκεί που λέγαμε όχι μόνο δημόσια κτίρια αλλά και ιδιωτικά κτίρια και ομάδες ιδιοκτητών ιδιωτικών κτίριων γιατί είχαμε τροπολογίες που επέκτηναν το πεδίο εφαρμογής όχι μόνο σε δημόσια κτίρια αλλά και σε τμήμα του ιδιωτικού τομέα. Κατόπιν συμφωνώ πλήρως με τους συναδέλφους για τους ρεαλιστικούς στόχους. Ε, αυτούς τους καιρούς, τους οικονομικά δύσκολους, της οικονομικής κρίσης, πρέπει να επιταχύνουμε τον κινητήρα της οικονομίας μας, δηλαδή τον τομέα της οικοδομής. Εάν επενδύσουμε στον τομέα των ακινήτων, επενδύουμε σε δουλειές και ταυτόχρονα σε θέσεις εργασίας. Είναι με κατάσταση αμοιβαία υποφελής, όπως αναφέρθηκε, και Μάλιστα, όπως είπαμε, το 20% είναι ρεαλιστικός ε, στόχος και δεν θα πρέπει να αναδιαπραγματευόμαστε το παρελθόν αλλά το μέλλον. Άρα... Συνεπώς θα έλεγα πρέπει να επιδιώξουμε τουλάχιστον το 20% και να το έχουμε ως δεσμευτικό στόχο. Τώρα όσον αφορά τα δεσμευτικά μέτρα, πιστεύω ότι είναι αυταπόδεικτο ότι είναι προτιμότερο να έχουμε δεσμευτικό στόχο παρά δεσμευτικά μέτρα. Εάν ωστόσο οι δεσμευτικοί στόχοι δεν είναι βέβαιοι, τότε θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε δεσμευτικά μέτρα. Πιστεύω ότι θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να τα συζητήσουμε και τα δύο. Κυρία Ποδηματά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, δύο παρατηρήσεις θέλω να κάνω, πολύ σύντομα. Πρώτα απ' όλα θέλω να υπενθυμίσω ότι βασικός στόχος της οδηγίας <clears throat> που συζητάμε είναι η ανάπτυξη και η ορίμανση αγορών στις ενεργειακές υπηρεσίες και στα αποδοτικά προϊόντα και με αυτή την έννοια θεωρώ ότι ο δημόσιος τομέας πρέπει να παίξει έναν ηγετικό ρόλο στην ε, προσπάθεια αυτή ε, στη διάρκεια της συζήτησης έγιναν πολλές παρατηρήσεις για το κόστος ε, και θέλω να επισημάνω ότι ουδής αμφισβητεί ότι το κόστος θα είναι ε, αρχικά υψηλό αλλά μεσοπρόθεσμα μέσω χαμηλότερων λογαριασμών για την ενέργεια μέσω της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας μέσω χαμηλότερων τιμών για τις ενεργειακές υπηρεσίες ε, είναι προφανές ότι τα ωφέλη θα γίνουν πολύ μεγαλύτερα και το αρχικό κόστος θα περιοριστεί. Ε, έγινε μεγάλη συζήτηση ε, για, την ικανότητα του δημόσιου τομέα να χρηματοδοτήσει φιλόδοξα μέτρα ιδίως σε περίοδο κρίσης και είναι προφανές ότι αυτές οι ανησυχίες είναι κατανοητές. Είμαι Ελληνίδα, κατανοώ και συμμερίζομαι απολύτως τις ανησυχίες αυτές. Πιστεύω όμως ότι υπάρχουν τρόποι να εξασφαλίσουμε ότι τα κράτη-μέλη ε, θα είναι σε θέση, επιλέγοντας έξυπνα μέτρα και έξυπνες πολιτικές, να αντεπεξέλθουν ε, στα φιλόδοξα αυτά μέτρα που προτείνονται στην οδηγία και υπάρχουν τροπολογίες που έχουν κατατεθεί και από μένα και από άλλους συναδέλφους προς την κατεύθυνση αυτή ε, και θέλω να αναφέρω ως παράδειγμα τις, τις ενεργειακές υπηρεσίες όπως οι συμβάσεις ενεργειακών επιδόσεων ε, που πιστεύω ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από δημόσιους φορείς γιατί ε, είναι ένα παράδειγμα γιατί προσφέρουν ε, αποτελεσματική λύση στο πρόβλημα των υψηλών αρχικών επενδύσεων για έργα βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας συνδυάζοντας το εγγυημένο κέρδος και τα ωφέλη πρόθεσμα. Για τη χρηματοδότηση, για τους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς που προτείνει ο εισηγητής ε, θέλω να επαναλάβω από την πλευρά μου ότι θεωρώ ότι είναι ζωτική σημασία ε, και είναι ζωτική σημασία γιατί μπορούν να δημιουργήσουν συνέργειες μεταξύ διάφορων διαθέσιμων ε, δημόσιων αλλά και ιδιωτικών πόρων και χρηματοδοτικών εργαλείων λαμβάνοντα λαμβάνοντας βεβαίως υπόψη και αυτό έχει τη σημασία του ότι σήμερα Ορισμένα κράτη-μέλη διαθέτουν εμπειρία σε αυτόν τον, ε, τομέα έχοντας ε, ήδη σε εφαρμογή παρόμοιους μηχανισμούς και άρα πρέπει να ε, εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα αυτού του είδους των μηχανισμών και των συνεργειών σε κάθε κράτος μέλος μέσω στήριξης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Τέλος, κύριε Πρόεδρε, οι ανησυχίες μας για το κόστος επίτευξης και αυτό είναι ένα γενικό συμπέρασμα της ενεργειακής αποδοτικότητας που είναι κατανοητές και θεμητές σε περίοδο κρίσης. Ε, πιστεύω ότι θα πρέπει να μας οθήσουν στο να αναζητήσουμε τους πιο αποτελεσματικούς και έξυπνους τρόπους ε, για να απαντήσουμε στα προβλήματα της χρηματοδότησης χωρίς να μας οδηγήσουν σε, ε, ε, στην επιλογή του να είμαστε λιγότερο φιλόδοξοι με δεδομένο ότι συμφωνούμε όλοι ότι τα ωφέλη της ενεργειακής αποδοτικότητας μέσω μακροπρόθεσμα ε, είναι πολλαπλά σε διάφορα επίπεδα και αφορούν όλους. Άρα νομίζω ότι ως, ε, Επιτροπή πρέπει να διατηρήσουμε τους, τους φιλόδοξους στόχους, μας, στόχους μας απέναντι σε ένα διστακτικό συμβούλιο και να ε, δώσουμε την εντολή στον εισηγητή και στους κοιόδης εισηγητές να ξεκινήσουν με μια ισχυρή εντολή διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο για δεσμευτικούς στόχους, αυτή είναι η βασική μου θέση, και αποτελεσματικά μέτρα για την επίτευξη των στόχων αυτών. Ευχαριστώ. Κλοντ, λοιπόν, ήθελε ε, να πει κάτι στο τέλο. Ε, έχετε το λόγο. Πόσο? Πιο δυνατά, δεν, ακούω. Ε, θα ήθελα τέσσερα λεπτάκια γιατί στην αρχή μίλησα λίγο. Ε, οι συνάδελφοι οι υπόλοιποι θα έχουν πρόβλημα μετά. Ε, εγώ είμαι εδώ πέρα μέχρι το τέλος συνεδρίασης, δεν έχω πρόβλημα. Αλλά υπάρχουν συνάδελφοι που έχουν και άλλα σημεία στη μερίσια διάταξη και θέλουν να μιλήσουν. Ε, σύντομα, σύντομα. Απλά μια παράκληση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Κέλλη ε, γιατί αφού πολλοί συνάδελφοι έθεσαν διάφορα προβλήματα, έθεσε την οδηγία σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Η οδηγία ενεργειακής αποτελεσματικότητας είναι νομοθεσία που μπορεί να βγάλει την Ευρώπη από την κρίση. Θα σας δώσω μόνο ένα νούμερο. Το 2011 το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου με την Ρωσία αυξήθηκε κατά άλλα 20 δισεκατομμύρια. Σήμερα έχουμε ένα έλλειμμα 77 δισεκατομμυρίων στο εμπορικό ισοζύγιο με τη Ρωσία. Δημιουργούμε λοιπόν πλούτο στην Ευρώπη και από αυτό το πλούτο στέλνουμε 77 δισεκατομμύρια στη Ρωσία. Σε ένα καθεστώς για το οποίο πολλοί από εμά έχουμε αμφιβολίες. Τι στόχο λοιπόν έχει αυτή η οδηγία. Να μείνει μέρος αυτού του πλούτου στο μέλλον στην Ευρώπη. Αυτό προσπαθούμε να επιτύχουμε. Και η Γερμανική Δημόσια Τράπεζα, η KfW, πριν από λίγες εβδομάδες ε, εξέδωσε την αξιολόγηση του 2010 για την ανακαίνιση κτηρίων. 9 ε, δισεκατομμύρια ε, επένδυσε το κράτος, 21 ε, δισεκατομμύρια ιδιώτες, 340.000 θέσεις εργασίας. Οπότε έρχεται το ερώτημα, ήταν αντικό αυτό για τον προπολογισμό. Το αποτέλεσμα της μελέτης είναι 1 ευρώ επενδύσεις σε ανακαίνιση έφερε 5 ευρώ στο γερμανικό προπολογισμό. Γιατί είχαμε λιγότερη ανεργία, περισσότερους φόρους και ΦΠΑ και τα λοιπά και τα λοιπά. Οπότε, συνάδελφοι, σταματήστε να το βλέπετε ως κάτι το οποίο είναι βάρος για την Ευρώπη. Αρχίστε να το βλέπετε ως μια ευκαιρία, γιατί όλες οι μελέτες μας δείχνουν πως όσο πιο αποτελεσματικοί είμαστε, τόσο ε, καλύτερα θα είναι η οικονομία μας. Και αυτό το οποίο άρα κάνουμε είναι να έχουμε, έχουμε την πολιτική απόφαση του 20% του Μαρτίου του 2007 που επαναλήφθηκε και το 2010 και 2011 από 27 αρχηγούς κρατών. Έχουμε αυτό το 20%. Ε, Μιλάμε λοιπόν για επιπρόσθετα μέτρα. Και αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι να σχεδιάσουμε αυτά τα μέτρα τα επιπλέον ε, έτσι ώστε να μπορούμε να τα λαμβάνουμε σε ολόκληρη την αλυσίδα της οικονομίας. Ένα σχόλιο για τα δεσμευτικά μέτρα και τους δεσμευτικούς στόχους. Εγώ συμφωνώ με την ε, μεταστροφή του ΕΛΚ που μέχρι τώρα ε, κατά πλειοψηφία τουλάχιστον ήταν κατά των δεσμευτικών στόχων. Νομίζω είναι θετικό το ότι επιτέλους καταλάβατε ότι χρειαζόμαστε δεσμευτικούς στόχους. Και όσο πιο δεσμευτικοί οι στόχοι, τόσο μεγαλύτερη η ασφάλεια για τους επενδυτές. Και νομίζω πως είναι πραγματικά θετικό. Αλλά ως διαπραγματευτική θέση πρέπει να πάμε με δεσμευτικούς στόχους και δεσμευτικά μέτρα. Γιατί όσοι από σας διαβάσετε το έγγραφο της Πολωνικής Προεδρίας θα καταλάβετε πως οι κυβερνήσεις ήδη με μεγάλη επιτυχία σχεδόν υποβάθμισαν τους στόχους και έχω την εντύπωση πως η Euroelectric και διάφορα άλλα λόμπι έρχονται σε εσά και σας λένε ξέρουν ήδη πως θα είναι δύσκολο να επιτύχουμε δεσμευτικούς στόχους στις διαπραγματεύσεις οπότε ξαφνικά πάνε, έρχονται σε εσά και λένε ε, δεσμευτικούς στόχους και ε, μετά δεν κάνετε τίποτα για τα μέτρα. Το είπα και την προηγούμενη φορά. Πρέπει να τελειώσουν οι διαπραγματεύσεις ε, με τρόπο ρεαλιστικό. Πρέπει να έχουμε την καλύτερη διατύπωση για τους στόχους και για τα μέτρα, αλλιώς δεν θα μπορέσουμε να παίξουμε τον ρόλο μας για να προχωρήσει αυτή η οδηγία. Έχω μόνο... Ε, δύο λόγια ακόμα για να απαντήσω συναδέλφους. Κρίμα, αλλά δεν φταίω εγώ. Φιώνα. Οι δημόσιες προμήθειες είναι κλειδί. Πρέπει να δούμε τη νέα πρόταση της Κομισιόν. Κύριε Πίπερ, ε, νομίζω πως ε, για το θέμα του ETS που αναφέρατε πρέπει να προσκαλέσουμε τον ε, συντάκτη της γνωμοδότησης της Επιτροπής Περιβάλλοντος και να συζητήσουμε μετά πώς έχουν τα πράγματα. Γενικά πρέπει να πω πως εάν δείτε την ψηφοφορία στην Επιτροπή Περιβάλλοντος υπήρχαν αρκετά προοδευτικές, ε, προοδευτικές συμβαστικές λύσεις από όλες τις ε, ομάδες. Ο Αλέχο έθιξε κάτι το οποίο είναι σημαντικό η διαχείριση της ζήτησης. Οπότε αυτή η οδηγία και το άρθρο 12 πρέπει να είναι πολύ ακριβή για να δημιουργηθεί κάτι το οποίο θα μειώσει το κόστος του ηλεκτρισμού στην Ευρώπη, κάτι το οποίο βεβαίως θα φέρει την ε, ορθή διαχείριση των κτηρίων και της βιομηχανικής παραγωγής στο παιχνίδι αυτό είναι καλύτερο αυτό από το να έχουμε παλιά αναποτελεσματικά εργοστάσια στη ΣΥΠΑ. Έχουμε εξοικονομήσεις ενός δισεκατομμυρίου σε κάποιες αγορές μέσω μόνο των μέτρων στην πλευρά της ζήτησης, οπότε θα πρέπει να κινηθούμε εδώ πέρα. Ε, λίγα τελευταία λόγια για το σύστημα των δημοσίων κτηρίων. Γνωρίζω πως ε, οι περισσότερες κυβερνήσεις έχουν δημοσιονομική κρίση. Γι' αυτό βεβαίως ε, το ανέφερε και η κυρία Γκροστέτ και η υπόλοιποι για την έννοια της ε, της εταιρεία η οποία εξοικονομεί ενέργεια. Ο Ρόναλντ Ρέιγκαν στη δεκαετία του 70 ε, είχε εισάγει την ανακαίνιση ε, την ανακαίνιση δημοσίων κτηρίων με τη Siemens, ABB και άλλες εταιρείες που μπήκαν στην αγορά αυτή. Οπότε πρέπει η αγορά αυτή να αναπτυχθεί τώρα που γνωρίζουμε πως ε, δεν μπορούν να ανταποκριθούν όλοι οι ε, προϋπολογισμοί. Αν θέλουμε στο μέλλον λοιπόν οι κυβερνήσεις να έχουν περισσότερα περιθώρια στον προϋπολογισμό δεν είναι καλό να μειωθούν κόστη των κτηρίων για να πάνε τα λεφτά αλλού, σε καινοτομία, για την υγεία, για άλλα ζητήματα, αλλά από αυτή τη σκοπιά δείτε, δείτε το κείμενο και δείτε πώς παλεύουμε για την ε, αγορά αυτή της ενέργειας στην Ευρώπη. Θέλουμε να απομακρύνουμε τα εμπόδια. Λοιπόν, την ερχόμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο, λόγω ε, των εκλογών που θα έχουμε θα έχουμε ίσως περισσότερο χρόνο από ό,τι σε άλλες εβδομάδες ολομελίες. Θα είμαι όλη την εβδομάδα στη διάθεσή σας. Όσοι συνάδελφοι έχουν λεπτομερείς ερωτήσεις, παρακαλώ, ελάτε σε επαφή μαζί μου να ανταλλάξουμε απόψεις ε, και ίσως, ε, κύριε Πρόεδρε, αν θα μπορούσατε να επιβεβαιώσετε πως με τις πέντε ε, συνεδριάσεις των σκιωδών εισηγητών που έχουμε προγραμματίσει ε, μπορούμε να έχουμε ως ε, στόχο να ψηφίσουμε 28 Φεβρουαρίου. Πρέπει να το δηλώσετε αυτό επισήμως για να ξέρουν όλοι οι συνάδελφοι τι θα γίνει τις επόμενες εβδομάδες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και για το ότι είσαι στη διάστηση των συναδέλφων για συζήτηση. Κατάλαβα πως η πρόταση είναι 28, 28 Φεβρουαρίου να ψηφίσουμε. Νομίζω λογικό αυτό, γιατί θα κερδίσουμε έτσι χρόνο. Προσωπικά αυτό το οποίο θα έλεγα είναι πως υπάρχει ο περιορισμός του να δούμε εγκαίρως της ε, συμβαστικές λύσεις. Θα πρέπει για να μπορέσουμε να ζητήσουμε και εναλλακτικέ λύσεις αν κάποιοι συνάδελφοι δεν είναι ικανοποιημένοι. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει ο καθένας να αποφασίσει μόνος του. Ε, τελειώνουμε λοιπόν με αυτό το σημείο και, το, και περνάμε στο επόμενο το οποίο είναι η COP17. Να σας παρακαλέσω να συνεννοηθούμε ο καθένας να μιλήσει μόνο δύο λεπτά. Ε, νομίζω μπορεί να μιλήσει μόνο αυτός ο οποίος θα μας ενημερώσει και να μην μιλήσουμε. Ε, κυρία Ντελκαστίγιο, λοιπόν, ξεκινάει. Είναι στο αυτά. Ντέρμαν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε που κάνετε και την εισαγωγή στο σημείο αυτό. Υπάρχει λίγη βαβούρα στην αίθουσα. Απόρρια της εργόδου συζήτησης που προηγήθηκε αλλά ήταν μια πολύ καλή συζήτηση. Λοιπόν, εν συντομία, σε σχέση με την συνάντηση του Durban, την λεγόμενη COP17, για τη δράση εναντί της κλιματικής αλλαγής. Σας παρακαλώ, αγαπητοί συνάδελφοι. Δυσκολεύεται το έργο με αναγκάζεται να μιλάω πολύ πιο δυνατά για να γίνω ακουστή. Αν μπορείτε να με βοηθήσετε θα ήταν πολύ καλό.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 Λίγα λεπτά για την κλιματική αλλαγή που έχει τόσο μεγάλη σχέση με την ενεργειακή αποδοτικότητα. Ησυχία παρακαλώ. Συνδέεται τα μάλα με το προηγούμενο θέμα το οποίο αντιμετωπίσαμε την τελευταία μία μισή ώρα. Λοιπόν, η διάσκεψη κορυφής του Durban, του Durban ήταν η συνάντηση παριθμών 17 σε σχέση με την κλιματική αλλαγή σε παγκόσμιο επίπεδο. Είχε το εξής αποτέλεσμα. Προς το παρόν, προς το παρόν. Μπορεί κανείς να δηλώσει ότι σε σχέση με το μέλλον των δράσεων για την κλιματική αλλαγή τα πράγματα είναι πιο ανοιχτά από ό,τι ποτέ. Από τη μία πλευρά έχει δημιουργηθεί μια πλατφόρμα, η λεγόμενη πλατφόρμα του Durban, όπου Καταρχήν υπάρχει συμφωνία να επιτύχουμε, να εφαρμόσουμε μια σειρά από μέτρα τα οποία δεσμεύονται να εφαρμόσουν όλα τα κράτη, τα οποία υπογράφουν αυτή τη συμφωνία. Από την άλλη πλευρά έχει παραταθεί η συμφωνία του Κιώτο με την απώλεια ορισμένων συμβαλωμένων μερών μέχρι το 2015 όπου θα δούμε τι, θα, τι μέτρα θα πρέπει να πάρουμε για το 2020, αλλά το πιο σημαντικό από τη δική μου άποψη είναι ότι αυτή τη στιγμή τα πάντα είναι ανοιχτά. Η πλατφόρμα του Durban δεν είναι παρά μόνο μια συμφωνία για το γεγονός ότι πρέπει να ξανασυμφωνήσουμε στο μέλλον. Αυτό είναι το συμπέρασμα. Από την άποψη αυτή λοιπόν πιστεύω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, η Κομισιόν, επικεφαλής αυτών, έχουμε μία ευκαιρία, έχουμε μία ανανεωμένη ευκαιρία να μπορέσουμε να θεσπίσουμε στόχους και τρόπους επίτευξης αυτών των στόχων που να είναι καινοτόμε και που να περιλαμβάνουν και περισσότερες χώρες, ιδίως τις χώρες που είναι οι μεγάλοι οι μεγάλε βιομηχανικέ χώρε οι οποίες εκπέμπουν αρία θερμοκηπίου. Ησυχία, λέει ο πρόεδρος. Πιστεύω λοιπόν ότι συνδεδεμένο με το θέμα αυτό της ενεργειακής απόδοσης ήταν και το θέμα της κλιματικής αλλαγής. Πρέπει λοιπόν να αντιμετωπίσουμε σωστά την ε, προοπτική μετά από τη διάσκεψη κορφής του Durban. Νομίζω ότι οι κοινοτικοί θεσμοί έχουν μία δυνατότητα να εκμεταλλευτούν αυτά τα νέα στοιχεία της πλατφόρμας του Durban για να μπορέσουν να εισαγάγουν νέες κοινέ προσεγγίσεις στο στόχο της επίτευξης της ενεργειακής απόδοσης. Τη στιγμή που απέχει ένα χρόνο περίπου η επόμενη συνεδρία για την κλιματική αλλαγή που θα γίνει στο Κατάρ, η Επιτροπή μας, και όχι μόνο η δική μας Επιτροπή, αλλά και η Επιτροπή Περιβάλλοντος, θα πρέπει να κάνουν τα απαραίτητα για να προχωρήσουμε προς την κατεύθυνση του να μπορούμε σε ένα χρόνο, μαζί με την Κομισιόν, να παρουσιάσουμε μια σειρά από δεσμευτικούς στόχους σε σχέση με την ενεργειακή απόδοση που θα πρέπει να σημαίνουν συγχρόνως και μια κοινή προσέγγιση μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης για τη μείωση των εκπομπών και να μπορέσουμε με αυτόν τον τρόπο να επιτύχουμε αυτό το οποίο δεν έχει γίνει πραγματικότητα μέχρι τώρα, να μπορέσουμε να ενσωματώσουμε αυτούς τους στόχους στο πρωτόκολλο του ΚΙΟΤΟ. Επομένω, η πρότασή μου είναι όταν έχουμε την ευκαιρία να μπορέσουμε να προχωρήσουμε προ την κατεύθυνση αυτή και ακριβώ μέσω των στόχων αυτών και των κοινών προσεγγίσεων για την ενεργειακή απόδοση να μπορέσουμε να προωθήσουμε αυτή, την, αυτή τη γραμμή πλεύσεως που νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα ελπιδοφόρα ιδίως αν συμπεριλαμβάνει και την απαραίτητη ευελιξία και τον απαραίτητο ρεαλισμό ελπίζουμε ότι με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε να πετύχουμε όλα αυτά τα οποία θέλουμε και να εκπληρώσουμε τους πόθους μας, βέβαια μετριάζοντας τους πόθους μας με τον ρεαλισμό για να μπορέσουμε να πετύχουμε αυτό το οποίο θέλουμε, να είμαστε αποτελεσματικοί. Παρά το γεγονός λοιπόν ότι δεν έχει επιτευχθεί πραγματικά τίποτα το καινοφανές στην συνεδρίαση του Durban σε σχέση με μια δεσμευτική συνθήκη, κάτι που κανένα δεν περίμενε ούτως ή άλλος. Παρ' όλα αυτά υπάρχει μια νέα διαφαινόμενη ευκαιρία και ένα θετικό στοιχείο, επειδή όλοι παραμένουν με ανοικτό πνεύμα και επειδή υπάρχει η αλλω παρ από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την Κομισιόν το Κοινοβούλιο να παίξουν ένα ηγετικό ρόλο σε σχέση με την περαιτέρω πορεία, εφόσον θα είμαστε σε θέση να εισαγάγουμε νέες καινοτομίες και νέες προόδους αυτό θα σημαίνει ότι έχουμε ένα ηγετικό ρόλο στα θέματα αυτά. Και θα ήθελα εν κατακλείδη να πω ότι αν καταφέρουμε να έχουμε μια κοινή προσέγγιση στους στόχους ενεργειακής απόδοσης, θα έχουμε πολλές δυνατότητες μπροστά μας. Ευχαριστώ. Thank you very much, Mr. Ευχαριστώ, κύριε Καστίγιο. Ευχαριστώ, κυρία Σίζελη. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να συμφωνήσω με την κυρία Ντελκαστήγιο. Ήταν μια πολιτική επιτυχία, αλλά και αυτοί οι οποίοι θέλαν βεβαίως κάτι το ουσιαστικό απογοητεύτηκαν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ πέρα ε, έπαιξε έναν ηγετικό ρόλο, ήταν επιτυχημένη. Θα ήθελα να συγχαρώ την ε, Επίτροπο για τις διαπραγματευτικές της ικανότητες. Αλλά αυτές οι διασκέψεις είναι μια καλή ευκαιρία να δούμε πώς, πού βρίσκεται το κάθε κράτος. Οι μεγαλύτερες χώρες, Κίνα, ΙΠΑ, Ρωσία, Γερμανία, Ιράν, Νότια Κορέα, Σαουδική Αραβία. Εκεί πέρα έχω την αίσθηση πως μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση ενδιαφέρεται να μειώσει τις εκπομπές και κανένας άλλος. Αυτό με ανησυχεί η κυρία Πιλάρ Καστίγιο. Ήδη μίλησε για το χρονοδιάγραμμα και την πλατφόρμα. Πρέπει να πω πως υπήρχαν και άλλα απτά αποτελέσματα, το ταμείο, η προσαρμογή του τεχνολογικού μηχανισμού, αλλά δεν μπόρεσε να περάσει ορισμένα πράγματα η Ευρωπαϊκή Ένωση όπω η μεγαλύτερη φιλοδοξία για τη μείωση των εκπομπών υπήρξε μόνο μια δέσμευση επί τη αρχής. Επίσης δεν υπήρξε ένα ενιαίος τρόπο υπολογισμού των εκπομπών, δεν υπήρξε πρόοδος ε, στην τομέα των αεροπορικών και των θαλάσσιων μεταφορών είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό να πούμε πως η διάσκεψη αυτή δεν έφερε τίποτα καινούριο στις υποχρεώσεις μείωσης των εκπομπών. Για εμάς είναι λοιπόν σημαντικό το σύστημα δέσμευσης και αποθήκευση άνθρακα να μπει στον μηχανισμό καθαρής ανάπτυξης. Και θα ήθελα να πω κάτι ακόμα. Θεωρώ πως εμείς ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προσπαθήσουμε να εφαρμόσουμε τις πολιτικές μας μέχρι το 2020 αν θέλουμε να συνεχίσουμε να παίζουμε ηγετικό ρόλο. Πρέπει να έχουμε επιτύχει τα ορόσημα μέχρι το 2020 και επίσης ε, ε, πιθανό είναι να πούμε πως η κλιματική αλλαγή αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία εξωτερικής πολιτικής για την Ένωση. Χρειαζόμαστε περισσότερη στήριξη. Είχαμε στήριξη από μικρότερες χώρες, ε, νησιωτικά κράτη. Αλλά... Άλλα κράτη δεν μας στήριξαν. Αυτό είναι μεγάλη πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και κάτι άλλο ακόμα όσον αφορά παραδείγματο χάρη ε, τον οδικό χάρτη στην Επιτροπή Ήτρε. Ε, δώσαμε τον ίδιο ρόλο με την Επιτροπή Ένβη. Αυτό θα πρέπει να γίνει νομίζω και να πάρουμε αυτό το ρόλο δηλαδή και για την κλιματική αλλαγή. Και εδώ πέρα ε, παίζει τον βασικό ρόλο η Επιτροπή Περιβάλλοντος. Όχι, πρέπει και εμείς να γίνουμε εδώ πέρα ισότιμοι εταίροι. Όπως τον Δεκέμβριο θα πρέπει να παίξουμε ισότιμο ρόλο και στο ψήφισμα. Εντάξει, συνεργαζόμαστε καλά με την Επιτροπή Περιβάλλοντος, αλλά εάν δείτε τον κατάλογο των μελών, ποιος έκανε τι, δεν, δεν το βλέπει αυτό και θεωρώ πως πρέπει να παίξουμε έναν ισότιμο ρόλο. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much, Mr. Ευχαριστώ πολύ κύριε Τσιζέλ για Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κατά την απόψη μου το αποτέλεσμα του Ντέρμπαν ήταν σημαντικό. Θα σας εξηγήσω γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε μια ατζέντα, ένα θεματολόγιο και αυτή συζητήθηκε καθ' όλη τη διάρκεια του κόπη. Είναι σημαντικό για την Ευρώπη το πιο σημαντικό όμως είναι ότι τα κυριότερα σημεία που προέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση εγκρίθηκαν. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα νοδικό χάρτη για όλ και τις 195 χώρες που συμφώνησαν σε αυτή την παγκόσμια συμφωνία, δηλαδή για τη συνέχιση του Τόκιο, του Κιώτο, και για τη δεύτερη δέσμευση του πρωτοκόλλου του Κιώτο. Έχουμε μια δεύτερη περίοδο δέσμευσης ε, έως ότου καταφέρουμε να επιτύχουμε παγκόσμια συμφωνία για τη παράταση του πρωτοκόλλου του Κιώτο και έχουμε μια βάση που ονομάζεται πλατφόρμα του Ντέρμπαν. Η πλατφόρμα του Ντέρμπαν είναι σημαντική διότι για πρώτη φορά όλες οι χώρες βρίσκονται σε ίδιο επίπεδο. Δεν υπάρχει διαχωρισμός αναπτυσσόμενων και βιομηχανοποιημένων χωρών ε, όπως είχε γίνει στην περίπτωση του πρωτοκόλλου του Κιώτο. Φυσικά διατηρείται η αρχή των διαφορετικών ευθυνών ε, ανάλογα με τις ικανότητες των διαφορετικών χωρών. Ωστόσο, όλες οι δεσμεύσεις θα είναι της ίδιας νομικής φύσης και όλες οι χώρες συμφώνησαν για αυτό. Αυτό θα αποτελέσει μια σημαντική βάση για να επεξεργαστούμε μια παγκόσμια συμφωνία. Το δεύτερο σημαντικό πράγμα της πλατφόρμας ε, του Durban είναι ότι υπάρχει ακόμα αρκετή αμφισημία. Αυτό σημαίνει ότι ίσως ε, εκπληρώσουμε αυτή τη συμφωνία με τα σημαντικά σημεία για την Ευρώπη. Για παράδειγμα, τη συμβατότητα της οικονομικής ανάπτυξης με την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και της φτώχειας. Υπάρχουν δηλαδή σημεία τα οποία θα χρειαστεί να συζητήσουμε και τα οποία είναι εξαιρετικά σημαντικά κυρίως για την δική μας επιτροπή όπως για παράδειγμα τι θα κάνουμε με τη βιομηχανία με τα βιομηχανικά μηχανήματα στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Συμφωνίας Καταπολέμησης Κλιματικής Αλλαγής το γεγονός ότι θα χρειαστεί να εστιάσουμε την προσοχή μας ε, και να λειτουργήσουμε σε ίσο επίπεδο με την Επιτροπή Περιβάλλοντος ώστε να παρέχουμε λύσεις ε, για αυτή την παγκόσμια συμφωνία. Και εδώ έχουμε χρόνο, διότι αυτό το, η δεύτερη περίοδος του Κιώτο θα μας δώσει το χρόνο να προετοιμάσουμε μια ικανοποιητική, ρεαλιστική ε, παγκόσμια συμφωνία που θα αντικαταστήσει το πρωτόκολλο του Κιώτο. Θα πρέπει λοιπόν να εμπλακούμε ενεργά από την αρχή και να συνεργαστούμε με την Επιτροπή Περιβάλλοντος ε, σε ίσο επίπεδο. Thank you. Ε, Ευχαριστώ. Ο, Επιτροπής ο κύριος Καρίδη, θα ήθελα τον λόγο. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Φυσικά συμφωνώ με όσα ακούσαμε. Το COP17 ήταν όντω μια διπλωματική επιτυχία. Το θεματολόγιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθοδηγεί πράγματι τη διαδικασία και κατά βάση επιτύχαμε όσα θέλαμε. Συμμερίζομαι λοιπόν όσα υπόθηκαν στις προηγούμενες ομιλίες. Επίσης καθίσταται σαφές ότι αυτή είναι μόνο η αφετηρία μιας μακροχρόνιας διαδικασία, η οποία θα διαρκέσει τουλάχιστον το 2015 όπου θα ολοκληρωθούν οι εργασίες ε, προετοιμασίας αυτής της νέας πλατφόρμας. Το 2015 η φετινή χρονιά θα είναι κρίσιμη διότι φέτος καθοριζόνται τα διαπραγματευτικά όρια αυτών των διαπραγματεύσεων και φυσικά ε, προσδοκούμε ε, να συνεργαστούμε με το ε, Κοινοβούλιο και με την παρούσα Επιτροπή για να καθοδηγήσουμε αυτή τη διαδικασία προς την κατεύθυνση που επιθυμεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Βλέπω πως ο κύριος Ρόιλ ξανάρχεται. Οπότε νομίζω πως θα παραδώσω την Προεδρία. Äh, Ευχαριστώ πάρα πολύ και περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Δεν δε βλέπω χωρίς γυαλιά. Äh, Κάρενς, έκθεση Κάρνς δηλαδή. Λοιπόν, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Διαμακρόν θα μιλήσω και λεπτομεριακώς γιατί είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση στην οποία προσβλέπω. Όχι, όχι, δεν θα μιλήσω για πολλή ώρα τότε. Καλά, δεν θα μιλήσω για πολλή ώρα. Όλοι έχουν διαβάσει τις προτάσεις μου. Είναι η δεύτερη ανταλλαγή απόψεων για αυτή την έκθεση. Αυτό το οποίο εγώ πιστεύω ότι είναι το πιο σημαντικό είναι από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να βοηθήσουμε να ενισχυθεί ο ρόλος της Κομισιόν σε ό,τι αφορά τον έλεγχο των διακυβερνητικών συμφωνιών, δηλαδή κυβερνήσεων μεταξύ της κυβερνήσεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παρόχων ενέργειας από τρίτες χώρες για να επιτύχουμε δύο αλληλένδετους στόχους. Ο πρώτος ο οποίος συνδέεται πάρα πολύ με αυτή την νομοθεσία είναι να εξασφαλίσουμε ότι οι συμφωνίες με τρίτες χώρες για την παροχή ενέργειας συμμορφώνονται με την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το τρίτο πακέτο λοιπόν για την ενέργεια θα πρέπει να εξασφαλίσουμε να πριτανεύει, να εξασφαλίζεται ότι δεν υπάρχει αποκλειστικότητα παροχή ενέργεια και οι καταναλωτέ μα έχουν τη δυνατότητα να έχουν τι καλύτερε δυνατέ τιμέ. Ο δεύτερο στόχο, και ο οποίο και αυτό απορρέει αυτή την νομοθεσία, είναι ότι όλα αυτά είναι ένα πρώτο βήμα για τη δημιουργία μιας εμβριακής κοινή Ευρωπαϊκή Φωνή στα ενεργειακά θέματα. Αν ενισχυθεί λοιπόν ο λόγο τη Ευρωπαϊκή Ένωση μεταξύ των διαπραγματεύσεων μεταξύ κρατών μελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση και παρόχων ενέργεια από τρίτε χώρε, σιγά σιγά θα αρχίζει να εισέρχεται σε αυτή τη διαδικασία ένα στοιχείο ε, κατά κάποιο τρόπο ομοιομορφίας θα μπορούσε να βοηθήσει τα κράτη-μέλη να έχουν βέλτιστες πρακτικές και να ενσωματώνουν αυτά τα στοιχεία Στι συμφωνίε αυτές, ώστε να υπάρχει προστασία των Ευρωπαίων καταναλωτών και να μπορούμε να απορρίπτουμε ορισμένε προτάσεις των κρατών μελών. Είναι σημαντικό λοιπόν η παρόχη ενέργειας από τις τρίτες χώρες, οι οποίοι δεν ενδιαφέρονται ιδιαίτερα στην νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντίθετα ενδιαφέρονται στην αποκλειστικότητα των συμφωνέων να κατανοήσουν την ανάγκη ανοιχτού ανταγωνισμού. Το να έχουμε λοιπόν τέτοιες ανοιχτές διαπραγματεύσεις, αυτό θα βοηθούσε τα κράτη-μέλη, είτε είναι μεγάλα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο ή μικρά, να έχουν μια καλή διαπραγμάτευση. Γιατί πολλές φορές όλοι μας είμαστε μικροί και κούτσικοι σε σχέση με μεγάλους παρόχους ενέργειας όπως είναι η Ρωσία που είναι ο μεγαλύτερος ουσιαστικά παραγωγός προμηθευτής φυσικού αερίου και πετρελαίου στον κόσμο. Με τον τρόπο αυτό λοιπόν θα έχουμε μεγαλύτερη δυνατότητα διαπραγματευτική για τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν διαπραγματεύονται με προμηθευτές από τρίτες χώρες ώστε να μην υπάρχουν ρήτρε αποκλειστικότητας γιατί με τον τρόπο αυτό αυτές οι ρήτρε θα μπορούσαν να αποτελέσουν αντικείμενο διαδικασίας παράβασης ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Οι δύο λοιπόν οι δυτοί αυτοί στόχοι είναι εξαιρετικά σημαντικοί σε αυτό το νομοθέτημα και οι προτάσεις οποίες εγώ έχω διατυπώσει είναι ότι προσπάθησα να διαγράψω πιο επακριβώς ποια θα έπρεπε να είναι η διαδικασία που θα υπησέλθει η Κομισιόν και εδώ θέλω να υπογραμμίσω δύο πράγματα. Καταρχήν είναι απαραίτητο να μπορέσει η Κομισιόν να συμμετέχει σε αυτές τις διαδικασίες σε πιο πρώιμο στάδιο. <clears throat> Αυτό θα έχει ενδιαφέρον και για τις εμπορικές εταιρείε οι οποίες είναι συμβαλόμενα μέρη γιατί αυτό θα αυξήσει την ασφάλεια δικαίου. Γνωρίζει κανείς ποιο είναι το πλαίσιο, είναι καλύτερο να ξέρει κανείς και να επενδύσει σε κάτι, ξέροντας ότι σε δύο-τρία χρόνια δεν θα ανατραπούν όλα αυτά και δεν θα βρεθεί ενώπιον μιας διαδικασίας επί παραβάση. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία της νομοθεσίας αυτής. Θα σταματήσω λοιπόν εδώ. Απλώς θέλω να σας υπενθυμίσω σε όλους ότι έχω ήρθει ήδη έρθει σε επαφή με όλους τους σκιώδεις εισηγητές, δύο φορές έχουμε συναντηθεί και φαίνεται ότι από την ε, χθεσινή μας συζήτηση ότι και οι άλλες πολιτικές ομάδες συμφωνούν με αυτή την προσέγγιση. Ας έχουμε ως τον πιο ενιαία στάση ώστε οι ενδεχόμενες αντιρρήσεις οι οποίες μπορούν να διατυπωθούν από την πλευρά του Συμβουλίου θα μπορέσουν να αντιμετωπιστούν με μια στεναρή και ενιαία στάση του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λάνια, να έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πράγματι, κύριε Σιγητά, σας ευχαριστώ για την προσέγγισή σας και την υποστηρίζω. Θεωρούμε όντως πως ο ρόλος ε, της Επιτροπής στον συντονισμό και την προώθηση της ε, συνεργασίας όσον αφορά τις εξωτερικές συμβάσεις ενέργειας πρέπει να ενισχυθεί έτσι ώστε αφενός να διασφαλίσουμε πως οι συμβάσεις θεύμα της κοινή ενεργειακής πολιτικής αναφερθήκατε στο πακέτο της εσωτερικής αγοράς, συζητάμε τον οδικό χάρτη 2050 και βεβαίως πρέπει να φροντίσουμε να ταιριάζουν στο πνεύμα αυτό και οι συμβάσεις αυτές και βεβαίως από την άλλη οι συμβάσεις αυτές έχουν πάντα επιδράσεις και σε άλλα κράτη-μέλη οπότε είναι μια κοινοτική υπόθεση που πρέπει να εξετάσει η Κομισιόν και υποστηρίζουμε την προσέγγιση του εισηγητού να γίνουν οι διαδικασίες πιο γρήγορες, πιο σαφείς για να έχουμε μια κοινοτική και σαφή πολιτική εδώ πέρα. Στις ε, συναντήσεις ε, με τους ε, σκιώδης ηγητές συνεννοηθήκαμε για κάποια πράγματα. Πρέπει νομίζω να ε, σκεφτούμε πως σε κάποιες τέτοιες συμβάσεις υπάρχουν και στοιχεία εμπορίου τα οποία περιέχονται προστασίας επενδύσεων και όταν διακυβεύονται αυτά τότε κινδυνεύουμε και εμείς γιατί βεβαίως ε, έχει συν, ε, αρμοδιότητα συνομοθέτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μετά την Λισαβόνα. Και άρα θα πρέπει εδώ πέρα να περιγραφεί επαρκώς ο ρόλος του Κοινοβουλίου και θεωρώ πως η Κομισιόν θα πρέπει σε τακτικά χρονικά διαστήματα, τακτά χρονικά διαστήματα να ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και για το τι έχει κάνει η Κομισιόν για να παίξουμε και εμείς τον ρόλο που μας αναλογεί. Αλλιώς θεωρώ πως έχει απόλυτο δίκιο ο εισηγητής πρέπει να είμαστε ενωμένοι και να εκπροσωπούμε τα κοινωτικά συμφέροντα. Σας ευχαριστώ. Ο συνάδελφος ο κ. Στόιρερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Για τους φιλελεύθερους θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την καλή συνεργασία να συνάδελφο ο κ. Μπέρντ Λάγκε ανέφερε τις πτυχές εμπορικής πολιτικής. Συμφωνούμε με αυτά. Βεβαίω θα μπορέσουμε ίσως να καταθέσουμε κάποιες ε, συμπληρώσεις στον τομέα της προστασίας των επενδύσεων, αλλά βεβαίω ταυτόχρονα είναι θέση μας πως σε όλη αυτή η υπόθεση δεν θα πρέπει να είναι πολύ γραφειοκρατική. Εμείς θεωρούμε πως ο ρόλος της Κομισιόν υπάρχει εκεί όπου τον ζητάνε τα κράτη-μέλη ζητάνε να δράσουμε από κοινού στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να διασφαλιστεί η ενεργειακή ε, ασφάλεια. Δεν θα πρέπει δηλαδή να υπάρξει κάποιο καταναγκασμός, αυτό πρέπει να το αποκλείσουμε και βεβαίως από την άλλη ε, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε πως ε, δεν θα πρέπει να ασχοληθεί με ιδιωτικές συμβάσεις η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά με διακρατικές ε, εκεί πέρα θεωρούμε πως υπάρχει ε, μία δυνατότητα παρέμβασης. Επίσης, ε, εκεί όπου υπάρχει εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχει ο ρόλος του Κοινοβουλίου, θεωρούμε πως ο δημοκρατικός έλεγχος θα πρέπει να ενισχυθεί σε όλους τους τομείς και αναζητούμε έναν τρόπο να ληφθεί υπόψη. Επαρκώς ο ρόλος του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Τζαβέλα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Καρίν για, μια, ε, για ένα κείμενο αρκετά δύσκολο. Ε, κύριε Πρόεδρε και κύριοι συνάδελφοι, έχω πολλά ερωτήματα όσον αφορά αυτή την ε, απόφαση την οποία καλούμεθα να πάρουμε. Ε, αυτό που βλέπουμε είναι ότι επιχειρείται ένας κεντρικός έλεγχος της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Αγοράς. Θεμητό. Μέσα στο κείμενο όμως της Επιτροπής αναφέρεται ότι επειδή η πρόταση αυτή έχει περιορισμένο, περιορισμένες οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις γι' αυτό δεν έγινε, δεν κρίθηκε αναγκαίο να γίνει μία μελέτη σκοπιμότητας τότε γιατί γίνεται. Για ποιο λόγο προχωρούμε σε αυτή την απόφαση. οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις δεν έχει, λέει το κείμενο της Επιτροπής. Γιατί προχωρούμε σε αυτή την κεντρική διαχείριση της ευρωπαϊκής ενεργειακής αγοράς. Προσωπικά δεν έχω αντίρρηση, έχω όμως κάποιες αντιρρήσεις σε κάποια από αυτά τα οποία επιχειρούνται με τις παρεμβάσεις οι οποίες επέρχονται. στείλουμε ένα μηχανισμό καταγραφής των διακρατικών συμφωνιών. Έως εδώ πολύ καλά. Το επόμενο βήμα είναι να δούμε αν αυτές οι διακρατικές συμφωνίες ακολουθούν την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Εξαιρετικά. Πράγματι και πρέπει να το κάνουμε. Ποια προβλήματα όμως δημιουργεί αυτή η παρέμβαση της Επιτροπής. Δημιουργεί προβλήματα στην εμπιστευτικότητα και στο απόρριτο των πληροφοριών όσον αφορά γεωπολιτική διάσταση του θέματος, δημιουργεί προβλήματα στην αγορά, έχοντας ένα χρονοδιάγραμμα αποφάσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο η αγορά δεν μπορεί να το περιμένει, και κάτι άλλο, κυρίες και κύριοι. Να ελέγξουμε την τήρηση των νομοθεσιών, ναι, της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Όταν όμως ζητούμε τήρηση των αποφάσεων των ευρωπαϊκών οργάνων, και θα μιλήσω πολύ συγκεκριμένα για να καταλάβουμε τι εννοώ. Οι αποφάσεις των ευρωπαϊκών οργάνων, παραδείγματος χάρη του Συμβουλίου, είναι ad hoc. Δημιουργείται κάτι και παίρνουν μια απόφαση. Έχουμε πίεση από τις Ηνωμένε Πολιτείε αυτή την περίοδο, επειδή είναι και προεκλογική περίοδο στην Αμερική, να προχωρήσουμε σε sanctions κατά του Ιράν. Υπάρχουν τέσσερις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία και η Ελλάδα, οι οποίες έχουν συμβάσεις προμήθειας Ιρανικού αερίου το Συμβούλιο παίρνει τις αποφάσεις για τα sanctions. Οι χώρες υπακούν και πράγματι διακόπτουν, αν μπορούν να διακόψουν κιόλα, αν είναι δυνατόν δηλαδή να εφαρμόσουν την ad hoc απόφαση του Συμβουλίου, διακόπτοντας την παροχή αερίου από το Ιράν. Τελειώνουν οι Αμερικανικές εκλογές και μετά από έξι μήνες οι Αμερικανοί κάπως τα βρίσκουν με τους Ιρανούς. Οι χώρες οι οποίες υλοποιήσανε την απόφαση του Συμβουλίου και μετά την παρέμβαση της Επιτροπής διακόψανε τη συνεργασία με το Ιράν, τι πρόκειται να κάνουν. Γι' αυτό θα έλεγα ότι σε αυτό το κείμενο, ναι, να έχουμε παρέμβαση. Αν τηρείται η ευρωπαϊκή νομοθεσία, πρέπει όμως να σκεφτούμε πώς θα δούμε την τήρηση των αποφάσεων των ευρωπαϊκών οργάνων όταν είναι ad hoc τρελαίνεται κάποιος ξέρω εγώ στο Ιράκ, ε, σκοτώνει κόσμο, παίρνουμε εμεί απόφαση, τι κάνουν. Όσοι έχουν συμβόλαια με το Ιράκ θα σταματήσουν αμέσως και απότομα η ενέργεια δεν είναι ένα προϊόν το οποίο μπορεί απότομα να κοπεί. Βλέπουμε επίσης στο κείμενο ότι ενώ είμαστε απόλυτοι για τις υποχρεώσεις των κρατών μελών εκεί όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει μεγάλο συμφέρον εξαιρούνται. Δηλαδή στο σημείο 5 του κειμένου βλέπουμε ότι διακρατικές συμφωνίες που γίνονται μεταξύ πολλών κρατών μελών κτλ. αυτές εξαιρούνται. Γιατί εξαιρούνται. Γιατί εδώ αναφέρεται μάλλον το κείμενο στο Σαχ Ντενής όπου το Ιράν επιτρέπεται κατ' εξαίρεση να συμμετέχει με 10%. Άρα έχουμε δύο μέτρα και δύο και στις εξαιρέσεις τις οποίες βλέπουμε εδώ. Και το τελευταίο το οποίο θα ήθελα να επισημάνω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προγραμματίζουμε ένα hearing για αυτό το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγματι αυτό το κείμενο. Σε αυτό το hearing, αυτό το οποίο βλέπουμε, είναι ότι έχουμε ομιλητές ή μάλλον προτιθέμεθα να έχουμε ομιλητές οι οποίοι δεν έχουν αντιρρήσεις πάνω σε αυτά που λέμε. Θα έλεγα κύριε Πρόεδρε ότι όταν έχουμε hearing θα πρέπει να φέρνουμε εδώ αυτούς οι οποίοι έχουν σοβαρότατες αντιρρήσεις σε αυτά τα οποία προτιθέμεθα να κάνουμε. Αυτή είναι η δημοκρατία και αυτός είναι δημοκρατικός διάλογος. Δηλαδή θα έπρεπε εφόσον η Ρωσία, καλός ή κακός, είναι ένας από τους κύριους προμηθευτές μας δεν θα έπρεπε στο, στο hearing να έχουμε επιδιώξει να έχουμε τη ρωσική πλευρά να δούμε πώς βλέπουν αυτοί αυτή την απόφαση την οποία προχωρούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, να σας πω μονάχα ότι για το θέμα της ακρόασης είχαμε κάνει μια συζήτηση μεταξύ των σκιωδών εισηγητών, των αρμοδίων ή των συντονιστών, συγγνώμη, συντονιστών θέλω να πω. Και τώρα έχουμε κάνει τις προκλήσεις, δεν μπορούμε να αλλάξουμε. Καταλαβαίνω αυτό που λέτε, έχετε δίκιο. Πρέπει πάντα στις ακροάσεις να καλούμε και αυτούς που έχουν αντίθετη άποψη. Αυτό έχει νόημα. Αλλά τώρα πια δεν μπορούμε να αλλάξουμε τις προκλήσεις. Και είναι τόσο μεγάλος και ο αριθμός των συμμετεχόντων που δεν έχει πια νόημα να κάνουμε κάτι τέτοιο. Κύριε Βιδάλ Κουάδρας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχουμε επιμείνει πολλές φορές ενώπιον της Κομισιόν ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει καλύτερος εσωτερικός συντονισμός μεταξύ κάτων μελών στα θέματα προμήθειας ενέργειας. Έχουμε κάνει προσπάθειες σε νομοθετικό επίπεδο για να δημιουργηθεί μια εσωτερική αγορά ενέργειας που να είναι πραγματικά ολοκληρωμένη. Και σε πολλούς τομείς της ενεργειακής πολιτικής έχουμε επιζητήσει τρόπους κοινή δράση. Και είναι προφανές ότι όταν πρόκειται για συμφωνίες με τρίτες χώρες και εκεί τα κράτη-μέλη είναι απαραίτητο να δείχνουν κάποιο στοιχειώδες πνεύμα αλληλεγγύης μεταξύ τους γιατί δεν θα μπορεί να είναι συμβατό με το πνεύμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ένα κράτος μέλος να συνάπτει συμφωνίες προμήθειας ενέργειας με μια τρίτη χώρα Προ το δικό του όφελο, αλλά συγχρόνω γνωρίζοντα ότι θέτει σε δυσκολότερη θέση τι άλλε χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε λοιπόν ένα μηχανισμό μετάδοση πληροφοριών, όπω προβλέπεται σε αυτό το νομοθέτημα, ώστε στι συμφωνίε μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών να υπάρχει ευρύτερη γνώση και πληροφόρηση. Ο συνάδελφός μας ο Κρίστιαν Κάριντς έχει παρουσιάσει μια έκθεση η οποία διευκρινίζει πολύ καλά την πρόταση της Κομισιόν και ε, καλύτερα σημεία τα οποία απαιτούν περισσότερη λεπτομεριακή αντιμετώπιση. Τι γίνεται όταν η Κομισιόν κάνει μια αξιολόγηση μια συμφωνίας αυτού του είδου μεταξύ μια χώρας και ενός τρίτου προμηθευτή. Τι συνέπειες θα πρέπει να προκύπτουν από αυτή την αξιολόγηση. Αν πρόκειται απλώ να κάνει μια αξιολόγηση και να μην, ε, να μην συμβεί τίποτα, τότε δεν έχει κανένα νόημα αυτό. Αυτό το οποίο προτείνει ο κύριος Κάνης είναι να προχωρήσουμε σε κάποιες περισσότερες διευκρινήσεις κρινήσεις στον τομέα αυτό και λέει ότι η αρνητική αξιολόγηση της Κομισιόν θα πρέπει να οδηγήσει σε μία όχληση προς το αρμόδιο κράτος μέλος και να του υποδειχθεί ότι αυτή η συμφωνία δεν συνάδει με το κοινοτικό δίκαιο και να αναφέρονται ακριβώς οι λόγοι αυτής της έλλειψης συμβατότητας. Το κράτη μέλος λοιπόν το οποίο τύχει αυτή τη προειδοποίηση και παρόλα αυτά συνάπτει αυτή τη συμφωνία θα πρέπει να ξέρει ότι η Κομισιόν μπορεί να κινήσει μια διαδικασία επί παραβάση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Πέραν τούτου υπάρχουν και δύο άλλα προεξάρχοντα στοιχεία. Πρώτα απ' όλα η ανάγκη να εξασφαλίσουμε ότι η ρήτρα εμπιστευτικότητας του άρθρου 7 να επεκταθεί σε κάθε πληροφορία που η Κομισιόν θα διαβιβάσει στα κράτη-μέλη. Άρα είναι απαραίτητο να υπενθυμίσουμε ότι αυτή η ρήτρα στα τρία εδάφια του άρθρου 3 να περιλαμβάνει αυτό το στοιχείο και αυτό θέλει να πτύχει ο κύριος Κράνης. Για να μην χρησιμοποιηθεί με καταχρηστικό τρόπο αυτή η ρήτρα εμπιστευτικότητος αναφέρει η έκθεση σαφώς τι ακριβώς θα πρέπει να έχει το χαρακτήρα εμπιστευτικών πληροφοριών. Και αυτό είναι μια μεγάλη επιτυχία του εισηγητή. Παρ' όλα αυτά είναι απαραίτητο να μην υπάρχουν επικαλύψεις στην κοινοποίηση αυτών των συμφωνιών προς την Κομισιόν και αυτό πολύ σωστά το έχει δει ο στην έκθεσή του στην αντίστοιχη τροπολογία βάσει της οποίας η κοινοποίηση η οποία παρουσιάζεται βάσει της πρότασης αυτής της απόφασης θα πρέπει να ακολουθεί αυτά που προβλέπονται στον κανονισμό ε, ασφάλειας εφοδιασμού, που εκεί ήμουν εγώ εισηγητής. Αυτό είναι μια πολύ θετική πτυχή λοιπόν της έκθεσης. Τέλος υπάρχουν και ορισμένε καινοτομίε οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές. Μία από αυτές είναι κάπως επικίνδυνη. Είναι εκεί που η Κομισιόν έχει το δικαίωμα να αξιολογήσει την συμμόρφωση με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όχι μόνο με, στα συμβόλαια τα οποία είναι υποσύναψη, αλλά και αυτά που έχουν ήδη συναυθεί. Εδώ όμως μπορούμε να μπούμε σε προβλήματα αναδρομικότητος της εφαρμογής του δικαίου. Αυτό είναι ολιστηρό έδαφος. Αλλά, παρόλα αυτά, κάποια από αυτά τα συμβόλαια έχουν μακρούς χρονικούς ορίζοντες. Εάν υπάρξει λοιπόν κάποια ε, κάποια δυνατότητα τροποποίηση ή μεταρρύθμισής του έχει καλώς. Αλλά το δικαίωμα, το, το στοιχείο της αναδρομικότητας είναι πολύ επικίνδυνο σε νομικό επίπεδο. Ένα άλλο στοιχείο είναι και το θέμα της εξάλληψης της πρόσβασης σε πληροφορίες που ένα κράτος μέλος έχει την υποχρέωση να δώσει στην Κομισιόν στην περίπτωση που προβλέπεται να γίνουν διαπραγματεύσει οι οποίε τροποποιούν μια υπάρχουσα συμφωνία ή οδηγούν σε μια νέα συμφωνία. Επομένω να μην υπάρχει πρόσβαση στα υπόλοιπα των υπόλοιπων κρατών μελών σε αυτές τις πληροφορίες υπό το πλαίσιο, μέσα στο πλαίσιο πάντα της ρήτρα εμπιστευτικότητας. Παρ' όλα αυτά μου φαίνεται μια πολύ καλή πρόταση και η έκθεση Currents βελτιώνει πάρα πολύ το κείμενο της Κομισιόν και γι' αυτό συγχαίρω τον εισηγητή. Ευχαριστώ, Hübner. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Μετά από όλα όσα υπόθηκαν, Ακόμη αναρωτιέμαι γιατί δεν έχουμε ε, τυποποιημένα σχέδια συμβάσεων. Εάν η Ένωση πρόκειται να συνάψει συμφωνίες με χώρες ε, ή ομάδες χωρών παροχής ενέργειας, γιατί να μην έχουμε μια τυποποιημένη φόρμα, ένα τυποποιημένο έντυπο. Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή είναι η κατάλληλη στιγμή. Αν θέλουμε να είναι ασφαλείς αυτές οι συμφωνίες, ε, να υπάρχει κάποιο είδου τυποποίηση, μια τυποποιημένη σύμβαση, την οποία θα εκπονήσει η Κομισιόν και μόνο σε εξαιρετικές περιστάσεις θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν διαφορετικές συμβάσεις ή διαφορετική διατύπωση. Το βασικό σκοπός φυσικά είναι ότι δεν θα πρέπει να υπάρχουν ε, νομικά ε, ή νομοθετικά λάθη σε αυτού του συμβάσει. Όπως είπε ο κ. Βινταλκουάδρο, θα μπορεί να υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία θα είναι εμπιστευτικά, ωστόσο το κυρίω κείμενο της ε, συμφωνίας θα μπορούσε να είναι τυποποιημένο. Δεν μιλάμε να δημιουργήσουμε κάποιο είδου τεχνητό ανταγωνισμό μεταξύ ε, χωρών που μας προμηθεύουν ενέργεια. Πρέπει απλά να διασφαλίσουμε την ενεργειακή μας ασφάλεια, την ε, ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού. Δεδομένου ότι χρειαζόμαστε ποικίλου ε, προμηθευτές. Ε, δεν συμφωνώ με την ιδέα πολλών εμπιστευτικών ε, και μυστικών διευθετήσεων. Θα ήθελα λοιπόν να ταχθώ υπέρ μιας τυποποιημένης σύμβασης η οποία θα έχει γίνει αποδεκτή από όλους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν θα έχουμε τέρμονες συζητήσεις με το κατά πόσο η συμφωνία είναι εντάξει κατά πόσο έχει άτυπες πτυχές ή τυπικές πτυχές. Πιστεύω ότι πρέπει να ξεφύγουμε από όλο αυτό. Στις οικοδομές, για παράδειγμα, έχουμε τυποποιημένες διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων και αυτές λειτουργούν μια χαρά. Με αυτόν μόνο τον τρόπο μπορούμε να διασφαλίσουμε σωστό θεμητό ανταγωνισμό και έτσι μπορούμε να ξεφύγουμε από όλες τις υποψίες και τις νομοσίες. Ποιος κάνει αν θέλει να απαντήσει. Ευχαριστώ πολύ για τα σχόλια. Πολύ χρήσιμα μου φαίνονται. Θα προσπαθήσω να απαντήσω συντομία σε κάποια από αυτά. Ε, πρώτα απ' όλα θα απαντήσω στην τελευταία ομιλήτρια, στην κυρία Χίμπνερ, για, την έλλειψη, για το να μην έχουμε αυτά τα σκοτεινά σημεία, σκοτεινές συμβάσεις, ε, παγίδες ή οτιδήποτε. Πρέπει να θυμόμαστε ότι υπάρχουν δύο επίπεδα συμβάσεων στην ενέργεια, οι διακυβερνητικές συμφωνίες, η IGA. Σε αυτές αναφέρεται αυτή εδώ η νομοθεσία και υπάρχουν οι εταιρικέ συμφωνίες, ε, ε, κάτι το οποίο δεν αφορά η παρούσα νομοθεσία. Στην πραγματικότητα οι περισσότερες συμφωνίες είναι εμπορικές στον τομέα της ενέργειας, είναι μεταξύ εταιριών ε, αυτές περιέχουν πληροφορίες με κόστο και διάφορες άλλες πληροφορίες που είναι εμπιστευτικές διότι οι εταιρείε που κερδίζουν χρήματα είναι και ευρωπαϊκές εταιρείε. Οποιαδήποτε εταιρεία εφόσον εάν δεν θα ήθελε να δημοσιοποιηθούν οι πληροφορίες εμπορικών συμφωνιών της, διότι θα βρισκόταν ε, σε μειονεκτική θέση σε σχέση με ανταγωνιστές που ενδεχομένως θα ήθελαν να υπογράψουν μια παρόμοια σύμβαση και θα μπορούσαν έτσι να προσφέρουν καλύτερους όρους. Πιστεύω ότι για οποιοδήποτε είδου σύμβαση, συμφωνία θα πρέπει να προστατεύσουμε την εμπιστευτικότητα των εμπορικών ευαίσθητων πληροφοριών. Ταυτόχρονα, επειδή εδώ μιλάμε για σημαντικές ενεργειακές συμβάσεις ε, που συχνά αφορούν πολλά έτη, τόσο οι ευρωπαϊκές εταιρείες καθώς και οι ξένοι ε, προμηθευτές ε, έχουν συμφέρον να υπάρχει στήριξη από κυβερνήσεις. Έτσι λοιπόν θα υπάρχουν αυτές οι διακυβερνητικές συμφωνίες που θα πρέπει να μελετώνται διεξοδικά. Ωστόσο αναφέρονται μόνο σε ορισμένες πτυχές αυτές οι συμφωνίες διακυβερνητικές των εμπορικών. Η Κομισιόν λοιπόν θα έχει ε, πρόσβαση σε πτυχές αυτές των IGA, των διακυβερνητικών συμφωνιών. Εφόσον ωστόσο το κρατό μέλη ορίσει αυτέ τι πληροφορίε ω εμπιστευτικέ, αυτέ τι πληροφορίε δεν θα πρέπει να κυκλοφορούν. Μιλάμε για μια κάπω ευαίσθητη διαδικασία εδώ πέρα. Προσπαθούμε να υπάρχει συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, θέλουμε να υπάρχει ομοιομορφία. Θα ήταν καταπληκτικό αυτό ως αποτέλεσμα αν χάρη στην ε, συμμετοχή της Κομισιόν υπήρχαν τυποποιημένες ρήτρε και όχι μόνο αυτό, αλλά και τυποποιημένε συμφωνίε που τα κράτη-μέλη θα μπορούσαν να χρησιμοποιούν ω βάση ε, και να υπάρχει απόλυτη συμμόρφωση με την νομοθεσία. Ωστόσο, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Καλό θα ήταν να μην παραβιάζουμε χωρίς λόγο το δικαίωμα εμπιστευτικότητα των εταιριών. Αυτό έχω γράψει μέσα στην προδοσή μου, νομίζω στο άρθρο 7, σε σχέση με την εμπιστευτικότητα αναφέρεται σαφώς. Ίσως κάποιοι να έχουν ιδέες το πώς θα μπορούσαμε να το κάνουμε ακόμη πιο αυστηρή αυτή τη ρήτρα, ότι δεν θέλουμε να παραβιάσουμε την εμπιστευτικότητα των εταιριών, θέλουμε να ανοίξουμε, ε, να, έχουμε, να είναι ελεύθερη η έρευνα στις ε, ε, διακυβερνητικές συμβάσεις αλλά το κομμάτι της συμφωνίας που θα αναφέρεται σε εμπιστευτικές εταιρικές πληροφορίες θέλουμε να διατηρείται εμπιστευτικό και οι πληροφορίες αυτές να προωθούνται μόνο στην Επιτροπή η οποία δεν θα το προωθεί στα υπόλοιπα κράτη-μέλη. Αυτά τα σχόλια είχα να πω επ' αυτού. Όσον αφορά το σχολείο της κυρίας Τζαβέλα, ειδικότερα όσον αφορά τις κυρώσεις για εταιρείε προμηθειών όπως του Ιράν, αυτή η νομοθεσία, όπως το βλέπω εγώ, δεν ε, αφορά αυτό το ζήτημα. Είναι παράπλευρη αυτή τη ζήτημα. Αυτό που λέει η παρούσα νομοθεσία είναι ότι εάν η Ελλάδα έχει μια συμφωνία με το Ιράν για προμήθεια ενέργειας ή επιθυμεί να υπογράψει ένα τέτοιο, μια τέτοια συμφωνία ή εαν η Βουλγαρία θέλει να υπογράψει κάτι τέτοιο με τη Ρωσία, ότι όλες αυτές οι διακυβερνητικές συμφωνίες θα πρέπει να συμμορφώνονται με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Ας υποθέσουμε ότι συμμορφώνονται υπάρχουν συμβάσεις της ε, Ελλάδας με είναι, τι συμμορφώνονται. Εάν το Συμβούλιο υιοθετήσει κυρώσεις που θέτουν σε κίνδυνο αυτή τη συμφωνία, ε, η κατάσταση θα είναι εξαιρετικά δύσκολη για την Ελλάδα ή για οποιονδήποτε έχει κάποια συμφωνία με το ΕΡΑΝ. Αυτή η νομοθεσία ωστόσο όπως και αν το ε, πάρουμε δεν, θα, δεν, απευθύνει, δεν αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα. Αυτό που λέμε είναι ότι πριν φτάσουμε στις κυρώσεις τι γίνεται με τις εναλλακτικέ ε, προμήθειες, ε, τι γίνεται εφόσον θέλουμε να διακόψουμε τη σύμβαση. Αλλά όλο αυτό είναι απόφαση του Συμβουλίου. Είναι κυβερνητική απόφαση. Δεν είναι νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, αφορά τη συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Είναι πολύ σημαντικό το ζήτημα που αναφέρεται. Αυτή η νομοθεσία όμως δεν αφορά αυτό το ζήτημα. Πρόκειται για απόφαση του Συμβουλίου. Δεν είναι, είναι νομοθεσία συμμόρφωσης ε, με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Well, I guess these are the only two... Αυτά είναι τα δύο σχόλια. Ε, νομίζω, α, υπήρχε και το ζήτημα του χρονοδιαγράμματος ε, οι εταιρείε ε, ανυπομονούν. Πιστεύω ότι αυτό θα είναι από τα πιο ε, δύσκολα ζητήματα. Έχω μιλήσει με διάφορους πολιτικούς για τα χρονοδιαγράμματα. Όπως κατάλαβα, κάποιοι στην Κομισιόν θα ήθελαν λίγο περισσότερο χρόνο για να προλάβουν να διαβάσουν όλες τις σελίδες. Κάποιοι στην Επιτροπή. Προτείνω εγώ σε περίπτωση που μια συμφωνία είναι εντάξει να έχουμε προθεσμία τουλάχιστον ε, το πολύ δύο μηνών όπου θα λαμβάνετε μια πράσινη καρτά από την ε, Κομισιόν ή τίποτα. Οι εταιρείε και ορισμένοι πολιτικοί θέλουν να είναι άμεσο. Ε, έχουμε και άλλους όμως που θέλουν να είναι ρεαλιστικό το έργο. Πρέπει να βρούμε μια μέση λύση. Κατά τα άλλα, σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ για όλες τις προτάσεις σας και αποτελεί πρώτη μου προτεραιότητα να ε, βρούμε προτάσεις ε, που η πλειοψηφία στην Επιτροπή θα συμφωνήσει. Χρειαζόμαστε ισχυρή, τονίζω, κοινοβουλευτική θέση, διότι στον, επόμενο, στον επερχόμενο τριμερή ε, διάλογο θα έχουμε να ξεπεράσουμε κάποιον σημαντικό ύφαλο και όσο περισσότερο ενωμένοι είμαστε, τόσο περισσότερη επιτυχία θα έχουμε. Ευχαριστώ, η κυρία Τζαβέλα. Κύριε ε, Καρέν, ευχαριστώ πολύ για τα σχόλια που κάνατε επί των σχολείων μου. Θα ήθελα να ήμουν πολύ συγκεκριμένη στα εκτιμώντας στην αιτιολογική σκέψη 2 λέει που συμμορφώνεται με, τον, με την νομοθεσία, με τις συνθήκες. Ναι, κάθε κράτος μέλος πρέπει να συμμορφώνεται με την νομοθεσία. Η αντίρρηση μου όμως είναι ότι όταν μιλάμε ότι πρέπει να συμμορφώνεται με τις πράξεις των θεσμικών οργάνων της Ένωσης, αυτές είναι πράξεις που λαμβάνονται ad hoc. Ενέργεια, πετρέλαιο και αέριο είναι αγαθά για τον κόσμο. Δεν μπορούμε να πούμε στην Ισπανία ότι το Συμβούλιο έλαβε μια απόφαση και ότι αυτό αποτελεί πράξη των ε, θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πώς πρέπει να σταματήσετε να εισαγάγετε ε, φυσικό αέριο και πετρέλαιο θα ήθελα να διαγραφεί η πρόταση resulting from the acts of the institutions of the union διότι εδώ μιλάμε για πράξεις που μπορεί να ληφθούν ad hoc και το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο δεν μπορεί να διακοπεί η, παροχή τους ad hoc και μετά να τα ξανανοίξουμε τις κάνουλες ε, συμφωνώ απόλυτα με τη συμμόρφωση ε, που λέτε με την ομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, αλλά τι θα γίνει με τις συμβάσεις αυτές με το Ιράν που είναι... και τι γίνεται με τη Γαλλία, την Ισπανία που, όπου υπάρχει μια σχέση προμήθειας με το Ιράν. Εντάξει, σύμφωνοι, θέλουμε να ασκήσουμε πίεση στο Ιράν, δεν έχω αντίρρηση γι' αυτό. Αλλά αν εμείς συμμορφωθούμε με αυτό και μετά γίνουν οι αμερικανικέ ε, εκλογέ. Σε έξι μήνε θα αλλάξουν τι σχέσει του με το Ιράν και τότε τι θα γίνει για τι υπόλοιπε χώρε. Και επίση στη διεθνή αγορά ε, θα ε, αυξηθεί σε τεράστιο βαθμό η τιμή του πετρελαίου και του αερίου. Γι' αυτό ζητώ να αφαιρεθεί αυτό το η πράξη των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Συμμόρφωση με την νομοθεσία βεβαίω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Να ρωτήσω την Κομισιόν αν θέλει να πει κάτι. Ναι, Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα σας. Ακούσαμε με μεγάλη προσοχή τις απόψεις που ε, εκφράστηκαν και είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι με το σχέδιο έκθεσης ε, ε, Κάρενς και αναμένουμε βεβαίω την τελική εκδοχή. Είμαστε ικανοποιημένοι για το ότι στηρίζει την γενική πρόθεση της Κομισιόν, τονίζει την ανάγκη να ενισχυθεί ο ρόλος της Κομισιόν και ξεκαθαρίζει πως ε, θα μπορούσε να αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα προς τη λεγόμενη ενιαία φωνή στις εξωτερικές συνεργειακές σχέσεις. Ε, να αναφέρω τρεις ε, τομείς που είναι ιδιαίτερα θετικοί στην έκθεση αυτή. Πρώτα απ' όλα την επιβεβαίωση πως υπάρχει μια κοινή αντίληψη του Γενικού Πεδίου Εφαρμογής Συμφωνίας και του ορισμού του τι αποτελεί διακυβερνητική ε, συμφωνία. Δεύτερον, επίσης θεωρούμε πως είναι σημαντικό να υπάρχει ανταλλαγή πληροφοριών και υποχρέωση ενημέρωσης κομισιών για μία έρευνα η οποία έχει ξεκινήσει ή θα ξεκινήσει. Κατόπιν επίσης σημειώνουμε την ε, παρουσία της Κομισιόν ως παρατηρητού στις ε, διακρατικές συμφωνίες και τρίτον προβλέπουμε έναν υποχρεωτικό ε, έλεγχο εξ άντε συμβατότητας όσον αφορά τη συμβατότητα με την ε, κοινωνική νομοθεσία. Να αναφέρω κάποια χαρακτηριστικά της πρώτης. Πρώτα απ' όλα δεν εμπλέκεται στην δυνατότητα των κρατών μελών να συνάψουν τέτοιες συμφωνίες. Είναι μόνο ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και της ε, Κομισιόν και υπάρχει επίσης βεβαίως και η υπηρεσία που παρέχει η Κομισιόν που είναι η αξιολόγηση της συμμόρφωσης. Οι υπηρεσίες Κομισιόν θεωρούν πως δεν υπάρχει ανάγκη ε, αξιολόγησης αντικτύπου. παρόλα αυτά κάναμε μια δημόσια διαβούλευση. Και οι οικονομικές ε, και κοινωνικές επιπτώσεις της πρότασης αυτής είναι έμεσες εάν ο μηχανισμός εφαρμοστεί οι επενδυτές έχουν μεγαλύτερη οικονομική βεβαιότητα και μετά η Κομισιόν μπορεί να διασφαλίσει πως το τρίτο πακέτο θα εφαρμοστεί προς όφελος των καταναλωτών, όπω τονίστηκε εδώ πέρα σήμερα. όπως είμαι σίγουρη ότι γνωρίζετε, η, συμβα... η εξελόγηση συμβατότητα ε, των διακυβερνητικών συμφωνιών είναι πολύ ευαίσθητο ζήτημα. Σε περίπτωση που μία υφιστάμενη συμφωνία αποσταλεί στην Κομισιόν και θεωρήσουμε πως δεν συμφωνεί με το κοινωτικό δίκαιο. Πρώτα απ' όλα η Κομισιόν στις περισσότερες περιπτώσεις θα έρθει σε επαφή με τα κράτη-μέλη να δει πώς μπορεί να επαναδιαπραγματευτεί ή ακυρωθεί η συμφωνία. Όσον αφορά τώρα το άρθρο 3 παράγραφος 1 θα ήθελα να σας πω πως κανονικά είναι πολύ ε, ευαίσθητο το ζήτημα του να δημοσιεύσει η Κομισιόν μια αξιολόγηση η οποία ομάθα λέει πως είναι ε, ε, ασύμβατη αυτή η συμφωνία. Μπορεί όμως να ξεκινήσει μια διαδικασία επί παραβάση και βεβαίω δεν προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις μια αξιολόγηση Κομισιόν και δεν θα προσθέσει και τίποτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ και εγώ. Να ανακοινώσω επίσης πως η προθεσμία για τις τροπολογίες είναι 17 Ιανουαρίου και περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης ασφάλεια ζωής το φυσικό κεφάλαιο στρατηγική 2020 και εδώ πέρα έχουμε την κυρία Σίσελη η οποία είναι η συγγήτρια έχετε τον λόγο Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε Μα ενδιαφέρει το θέμα της στρατηγική, η στρατηγική διατήρησης της βιοπικιλότητας και του φυσικού, των φυσικών πόρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρετε το έτος του 2010 ήταν το έτος βιοπικιλότητος και έλαβε χώρα και με μια μεγάλη διάσκεψη για τη βιοπικιλότητα στην Αγκόγια, στην Ιαπωνία και καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι από το 2010 μέχρι το 2020 θα πρέπει να έχουμε τη δεκαετία της διατήρησης της βιοπικιλότητας. Ωραία και μεγάλα λόγια. Η πραγματικότητα όμως είναι πολύ διαφορετική. Βλέπουμε ότι κατά 25% των, τα είδη των ειδών στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υποκίνδυνο εξαφάνισης 90% των ηχθείων που αλλιεύουμε επίση βρίσκονται σε κίνδυνο εξαφάνιση βάσει των μελετών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Κάθε χρόνο χάνεται το 3% της, ε, των ειδών που βρίσκονται σε παγκόσμιο επίπεδο λόγω της απώλειας βιοπικιλότητος. Νομίζω λοιπόν ότι είναι απαραίτητο να σκεφτούμε καλύτερα για μια στρατηγική προστασία της βιοπικιλότητος στον ε, ορίζοντα του 2020 θα πρέπει να προβλέψουμε τις αντίστοιχες χρηματοδοτήσεις και τις πολιτικές κατευθύνσεις σε οριζόντιο επίπεδο. Πιστεύω ότι είναι και ο κατάλληλος χρόνος να πράξουμε κάτι έναντι της απώλειας βιοπικιλότητας. Η πρόταση αυτής της Κομισιόν συμπεριλαμβάνει και μια συνολική ένα συνολικό όραμα για την προστασία των βιοτόπων μέχρι το 2020. Είναι απαραίτητο η Κομισιόν να έχει καταθέσει προτάσεις για τα θέματα αυτά, τους στόχους της μαζί με τα απαραίτητα συνοδευτικά μέτρα και οι στόχοι αυτοί είναι να μπορέσουν να επανέλθουν στη φυσική τους κατάσταση τα ενδιατήματα και οι φυσικοί βιότοποι ώστε να προστατευτούν τα ίδια αυτά, να υπάρξουν περιορισμοί για τις γεωργικές δραστηριότητες και στο επίπεδο της αλίας, ο πέμπτος από τους έξι στόχους της Κομισιόν. Περιλαμβάνει τον αγώνα εναντίον ε, παρήσακτων ειδών τα οποία μπαίνουν στους φυσικούς αυτούς βιοτόπους και επίσης προβλέπεται μια μεγαλύτερη συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία της βιοποικιλότητας. Κατά την άποψή μου λοιπόν και το αυτό αντανακλάται και στη γνωμοδότηση που έχω προετοιμάσει για την Επιτροπή μας κάτι το οποίο μου φάνηκε εμένα πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι η η απώλεια βιοπικιλότητος οδηγούν και σε απώλεια ουσιαστικά εθνικού προϊόντος στις χώρες μας. Αν χάσουμε τη βιοπικιλότητα αυτό έχει και κάποιο αντίκτυπο στο επίπεδο της ευμαριάς μας. Ένα δεύτερο στοιχείο είναι ότι η βιοπικιλότητα δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί μονάχα με επιμέρους πολιτικές, αλλά θα πρέπει να ενσωματωθεί σε όλες τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τρίτον, ότι η, σας υπενθυμίζω ότι η Κομισιόν είχε ανακοινώσει μια στρατηγική για τις πράσινες υποδομές μέχρι το 2012. Ξέρουμε ότι η Κομισιόν δεν εκπλήρει πάντα τα χρονοδιαγράμματα τα οποία θέτει, πολλές φορές καθυστερεί, αλλά το πλαίσιο αυτό δεν είναι αρκετά φιλόδοξο. Θα πρέπει αυτή η στρατηγική το ταχύτερο δυνατόν να εκπονηθεί. Χρειαζόμαστε και καλύτερη συνέργεια μεταξύ των πολιτικών που εμείς προετοιμάζουμε. Έχουμε τις προτάσεις κομισιών για τις υποδομές ε, μεταφορών, ενέργειας, ε, περιβάλλοντος. Θα πρέπει να έχουμε λοιπόν μια πιο πράσινη υποδομή το ταχύτερο δυνατό. Και ένα άλλο στοιχείο είναι το να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στην γνώση, στην καινοτομία και την έρευνα στον τομέα αυτό. Δεν χρειαζόμαστε μονάχα την επιστημονική γνώση για να αξιολογήσουμε καλύτερα την κατάσταση. Χρειάζεται να μας δώσει η επιστημονική εμπειρογνωμοσύνη και καλύτερη γνώση για τη διάδραση μεταξύ των διαφόρων φυσικών ειδών και για τον καλύτερο, το τρόπο προστασίας της βιοποικιλότητος. θα πρέπει να κατανοήσουμε την αξία που περιέχει η βιοπικιλότητα για τα προϊόντα μας και τις διεργασίες μας. Γι' αυτό η απώλεια βιοπικιλότητας εξακολουθεί να αποτελεί ένα μεγάλο πρόβλημα για τις κοινωνίες μας. Και θα πρέπει να υπάρξει και η εσωτερικοποίηση του εξωτερικού κόστους που προέρχεται από την απώλεια της βιοπικιλότητας. Και αν δεν το πράξουμε αυτό, δεν μπορούμε να διατηρήσουμε εποφελώς τη βιοπικιλότητα. Όλα πρέπει να έχουν και κάποιο τίμημα ώστε να μπορεί να ενσωματώνεται το κόστος τους. Είναι απαραίτητο επίσης να εξασφαλίσουμε και καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών μέσα στα πλαίσια των πολιτικών που ασκούνται για την προστασία της βιοπικιλότητας και αυτό είναι απαραίτητο ιδίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν ένα ζωτικό συμφέρον να εξασφαλιστεί αυτή η παροχή πληροφοριών, δεν μπορούν να αποκομίσουν από μόνες τους τις πληροφορίες, να κάνουν δικές τους μελέτες Γι' αυτό θα πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να έχουν με την ανταλλαγή πληροφοριών και την μεταλαμπάδευσή του τα απαραίτητα στοιχεία για τη δραστηριότητα, δραστηριότητά τους. Και εν κατακλείδη θα ήθελα να σας υπενθυμίσω και τη σχέση βιοπικιλότητας και κλιματικής αλλαγής. Είναι απαραίτητη η εφαρμογή όλων των πολιτικών που έχουμε στον τομέα του περιβάλλοντος, γιατί ακριβώς ο τομέας του περιβάλλοντος είναι αυτός όπου καθυστερεί πολύ η εφαρμογή των κοινοτικών μέτρων. Η προθεσμία για τις τροπολογίες μέχρι τις 16 Ιανουαρίου και στις 6 Φεβρουαρίου θα γίνει ψηφοφορία στην Επιτροπή μας. Ευχαριστώ. Αυτά από τη δική μου πλευρά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, η προθεσμία για τροπολογίες είναι γνωστή. Η Κομισιόν θέλει να πει κάτι. Ναι. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω για το ζήτημα της βιοποικιλότητας και να αναφέρω κάποιες ε, ξεκαθαρές απόψεις για τη στρατηγική και βλέπουμε έτσι μια ευθυγράμμιση που υπάρχει και ενίσχυση της εφαρμογής ε, της στρατηγικής που στηρίζεται και από όλους τους κλάδους όπως ανέφερε και η συγκέτρια είναι κάτι το απαραίτητο για την επιτυχία αυτής της στρατηγικής θα ήθελα να Είμαστε σίγουροι πως όλοι είμαστε έτοιμοι για αυτή τη στρατηγική και για μια επιτυχή εφαρμογή η οποία θα εξαρτηθεί στην κοινή, από την κοινή μας προσπάθεια για να εφαρμόσουμε τα υπεσχημένα. Σας ευχαριστώ λοιπόν για τις απόψεις σας και για τη δουλειά που έχετε κάνει για να ενσωματώσετε τη βιοπικιλότητα στις άλλες τομιακές πολιτικές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, 17 Ιανουαρίου, το επαναλαμβάνω, οι τροπολογίε. Τελειώσαμε με αυτό το σημείο τη ημερήσια διάταξη. Οι σκιώδει συγητές δυστυχώ λείπουν όλοι. Και περνάμε απευθεία στο επόμενο θέμα, το υπαριθμόν 7. Ασφάλεια τροφίμων για τρόφιμα για μικρά παιδιά και τρόφιμα με ειδικού ιατρικού σκοπού. Εδώ πέρα ο κύριος Τάκουλα είναι ο συγητής και του δίνω το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αυτό όπως είπατε αφορά τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς και για βρέφη και μικρά παιδιά. Δίνουμε μια γνωμοδότηση, υπάρχει μια γνωμοδότηση εδώ ε, προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος. Στη γνωμοδότηση αυτή ε, την εξέτασα ε, από την άψη της βιομηχανίας, ε, ε, της ενέργειας, της έρευνας και της καινοτομίας. Το ζήτημα είναι αρκετά τεχνικής φύσης. Ίσως αναρωτηθείτε για ορισμένες από τις πτυχές, ειδικότερα αυτές που περιλαμβάνει διάφορες μορφές ε, ε, τροφίμων για βρέφη και μικρά παιδιά όπως, δημητριακά, όπως ε, παιδικά τρόφιμα που βασίζονται σε δημητριακά και ούτω καθεξής. Και επομένως δεν περιλαμβάνει όλα αυτά τα τρόφιμα των κατηγοριών αυτών. Πρόκειται για προϊόντα για διαβητικούς και για τα προϊόντα για αθλητές. Η Κομισιόν λοιπόν σε διάφορα οριζόντια κείμενα αντιμετωπίζει, λέει ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν ιδιαίτερα αυτά τα, αυτά τα προϊόντα, αυτά τα τροφιμικά προϊόντα. Η πρόταση λοιπόν της Κομισιόν αναφέρει ότι τα διαιτητικά τρόφιμα δεν πρέπει να περιληφθούν εδώ, αλλά εγώ νομίζω ότι και για αυτά τα τρόφιμα θα πρέπει να λεχθεί κάτι στην έκθεση αυτή. για αυτά τα προϊόντα τα οποία προβλέπονται ως ε, τα οποία, πρέπει να, τα οποία μπορούν να λαμβάνονται με το σκοπό της μείωσης του βάρους από τα άτομα για ένα χρονικό διάστημα. Υπάρχουν όμως συγκεκριμένοι κανόνες για την ε, ετικετοθεσία στα προϊόντα τα οποία δεν περιέχουν γλουτένη. Ήδη η Κομισιόν έχει υποβάλει προτάσεις προς την κατεύθυνση αυτή. Μετά όμως τις συζητήσεις με διάφορους συναδέλφους, εγώ έχω καταλήξει στο συμπέρασμα ότι εδώ η Επιτροπή Περιβάλλοντος θα πρέπει να θέσει προτάσεις για αυτά τα θέματα γιατί αυτή είναι η αρμόδια επί της ύλης. Αυτοί λοιπόν έχουν τη βασική ευθύνη. Εμείς θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας στα θέματα στα οποία έχουμε πραγματική αρμοδιότητα. Επομένως, παρά το γεγονός ότι όλα αυτά τα στοιχεία είναι ιδιαίτερα τεχνικά, δεν πρόκειται για ένα καινοτόμο θέμα, κάτι το οποίο είναι καινούριο, και έχουμε καταφέρει να καταλήξουμε σε ένα κοινό πλαίσιο και κατά συνέπεια μπορώ να σας πω ότι οι προτινόμενες τεχνικές ε, τροποποίησεις μπορούν να συμπεριληφθούν στο κείμενο τους της πρότασης. Και επίσης εγώ προσωπικά έχω καταθέσει μια σειρά τροπολογιών και τρέχει η προθεσμία καταθέσεως και μέχρι την Τρίτη. Ίσως μπορώ να κλείσω εδώ στο σημείο αυτό και αν θέλουν να πούν κάτι οι συνάδελφοι είμαι έτοιμο να τα αντιμετωπίσω τα σχόλιά τους. Ευχαριστώ πολύ κυρία Γκρος Τέντ. Έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα ήθελα να πω ότι εδώ μιλάμε για ένα θέμα εξαιρετικά σημαντικό. Σημαντικό διότι αφορά την προστασία των καταναλωτών και ταυτόχρονα την καινοτομία καθώς και την προσοχή που δίνουμε στην ε, διατροφική βιομηχανία, σας υπενθυμίζω βιομηχανία που έχει τις ε, πολύ ψηλές εισαγωγές ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η αγροδιατροφική βιομηχανία λοιπόν χρειάζεται την υποστήριξή μας καθώς ερευνά την προσαρμογή των τροφίμων για συγκεκριμένες ομάδες καταναλωτών, ομάδες στόχους καταναλωτών, είτε πρόκειται για βρέφη, θα μιλήσω και για αυτά, είτε πρόκειται για αθλητές, είτε πρόκειται για άτομα με δυσανεξία στη γλουτένη, στη λακτόζη και ούτω καθεξής, είτε πρόκειται για ένα άλλο πολύ συχνό φαινόμενο άνθρωποι που θέλουν να χάσουν βάρος. Είναι πολύ σημαντική λοιπόν αυτή η έκθεση, αυτή η πρόταση κανονισμού. Είναι θεμελιώδους σημασίας και αφορά όλους τους συμπολίτε μας σε κάποια στιγμή της ζωής τους. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να μελετήσουμε διεξοδικά αυτό το ζήτημα. Ε, ε, συμμερίζομαι το σκεπτικό του ε, εισηγητή, του κύριο Τακούλα. Είναι πιο δύσκολο τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τις αρχές ελέγχου να ξεχωρίσουν τα τρόφιμα που απευθύνονται στο γενικότερο πληθυσμό και τα τρόφιμα που απευθύνονται στις συγκεκριμένες ομάδες που ανέφερα επιβάλλεται να διατηρήσουμε υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών για αυτά τα συγκεκριμένα τρόφιμα διότι εδώ μιλάμε για διατροφική ασφάλεια αλλά και για προστασία της υγείας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί να διευκολύνει τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς απλοποιώντας την νομοθεσία και περιορίζοντας το διοικητικό άκθος. Εκεί συμφωνούμε με την Κομισιόν. Υπενθυμίζω επίση, και τώρα απευθύνομαι στην Κομισιόν ότι όλο αυτό δεν πρέπει να γίνει ει βάρο της προστασίας των καταναλωτών. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε μια σωστή ισορροπία μεταξύ των δύο. Έχουμε κατηγορίε προϊόντων που καλύπτονταν από την προηγούμενη οδηγία και που σήμερα έχουν εξαιρεθεί από την πρόταση τη ε, Κομισιόν. Έτσι συντομεύουμε τις υπαρξές διατάξεις όσον αφορά τις προτάσεις και τη σήμανση, τις ετικέτες και αυτό μπορεί να θέσει προβλήματα διότι η εγκατάλειψη ορισμένων κριτηρίων ε, σύνθεσης ή κάποιων όρων σήμανσης μπορεί να επιφέρει κινδύνους για τον ελλιπώς ενημερωμένο καταναλωτή. Όσον αφορά τα τρόφιμα χαμηλής θερμιδικής περιεκτικότητας που απευθύνονται σε όλο και περισσότερους ε, καταναλωτές που θέλουν να χάσουν βάρος γιατί αυτό είναι και της μόδας. Η κατανάλωση αυτού του είδους τροφίμων απαιτεί συνήθως ιατρική συμβουλή, ιατρική παρακολούθηση. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να έχουμε ένα συγκεκριμένο κείμενο το οποίο να αφορά αυτή την ομάδα διότι υπάρχει κίνδυνος κάποιες επιχειρήσεις, κάποιοι βιομηχανοί οι οποίοι ορισμένοι από αυτούς θα είναι πολύ σοβαροί και θα συνεχίσουν να παρέχουν όλες τις πληροφορίες σε σχέση με το προϊόν που προτείνουν σε αυτές τις συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού αλλά κάποιοι άλλοι βιομηχανοί λιγότερο σοβαροί θα πούν ας υποφεληθούμε από την ομοθεσία λέγοντας ότι ναι αυτό το προϊόν είναι καλό προϊόν για όσους θέλουν να χάσουν βάρος χωρίς ε, να υπάρχει ο ίδιος έλεγχος και η διαυστηρότητα. Αυτό που λέγω λοιπόν είναι ότι πρέπει να προσέχουμε πολύ διότι έχουμε, έχουμε μεσαίες επιχειρήσεις που παράγουν συγκεκριμένα ε, προϊόντα και οι οποίες μπορεί να υποστούν τον ανταγωνισμό από μεγάλες επιχειρήσεις. Ε, για παράδειγμα με τους Ολυμπιακούς Αγώνες η Coca-Cola θα βγάλει ένα προϊόν το οποίο όπως φαίνεται ε, σύμφωνα με τις διαφημίσεις θα είναι ιδανικό ε, για την αντοχή των αθλητών. Ξέρουμε πολύ καλά ότι η Coca-Cola δεν είναι και η πιο κατάλληλη για να προτείνει ε, ένα προϊόν το οποίο θα βοηθάει στη διατήρηση της αντοχής των αθλητών. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Φοβάμαι ότι αν αφαιρέσουμε ορισμένα, αν δεν συμπεριλάβουμε κάποια από αυτά τα προϊόντα σε αυτόν τον κανονισμό, αυτό θα προκαλέσει σύγχυση στους καταναλωτές αλλά και αθέμητο ανταγωνισμό για τις βιομηχανίες. Γι' αυτό είμαι λίγο ανήσυχη. Θα ήθελα λοιπόν να προσέξουμε. Επίσης και το ζήτημα των τροφίμων χωρίς γλουτένη και μίλησε γι' αυτό ο εισηγητής μας. Και εκεί η μόνη θεραπεία που υπάρχει για αυτά τα άτομα οι οποίοι είναι ασθενείς έτσι δεν έχουν τις ανεξίες στη γλουτένη είναι άτομα για τα οποία πρέπει να ανησυχούμε διότι διότι εάν δεν μπορούν να έχουν στη διάθεσή τους τα πολύ συγκεκριμένα προϊόντα που χρειάζονται μπορεί να υπάρχουν δυσάρεστες ε, επιπτώσεις. Επίσης θα ήθελα να μιλήσω τώρα για το γάλα ανάπτυξης το οποίο περιορίζουμε στο, στο ένα έτος και μετά από ένα έως τρία λέμε α, δεν ασχολούμαστε πλέον με αυτό τότε μπορούμε να δώσουμε οποιοδήποτε τύπο γάλακτος Λυπάμαι όμω ε, από ηλικία ενός έω τριών ετών πρέπει να προφυλάσσουμε το παιδί διότι μπορεί να υπάρχουν ε, ζυζανιοκτόνε μέσα σε αυτό το γάλα το οποίο θα δώσουμε σε ένα παιδί που είναι ηλικία ενός έω τριών ετών. Γιατί να προσέξουμε δηλαδή ένα βρέφο ηλικία μέχρι ενός έτου και αφού ε, κλείσει το ένα έτος δεν έχει πια το δικαίωμα να προστατευτεί με τον ίδιο τρόπο θα ήθελα λοιπόν εγώ να συμπεριλάβουμε τα γαλακτοκομικά προϊόντα που απευθύνονται σε παιδιά έως ηλικία τριών ετών γιατί πιστεύω ότι και αυτή η κατηγορία είναι σημαντική. Όπως έχουν τα πράγματα σήμερα, η πρόταση προβλέπει αυτές τις εξαιρεσει ε, Αυτό αυτού του καλού. Πιστεύω ότι ο κίνδυνος είναι μεγάλος. Δεν πρέπει να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ την προσοχή λοιπόν της Κομισιόν για αυτό το θέμα. Στη συνέχεια, έχω μιλήσει ήδη για τα προϊόντα διατροφής για αθλητές, δεν θα επανέλθω. Αυτό που είναι σημαντικό στα εκτιμώντας 3 και 29, ο εισηγητής αναφέρεται στο ζήτημα της έρευνας και της καινοτομίας στον τομέα της διατροφής. Πρέπει να επιτραπεί η διάθεση στην αγορά γρήγορη τροφίμων που, που προορίζονται για συγκεκριμένη διατροφή και που προέρχονται από επιστημονική έρευνα. Όλοι συμφωνούμε σε αυτό. Συμμερίζομαι επίση με τι συστάσει του εισηγητή που θέλει να ενισχύσει τι ανεξάρτητε επιστημονικέ αξιολογήσει για τα τρόφιμα που είναι καταλληλότερα για τις διατροφικές ανάγκες συγκεκριμένων πληθυσμών συμφωνούμε με αυτό, στη γνωμοδότηση της Επιτροπής ΙΤΡΕ πρέπει να ενισχύσουμε τη νομική ασφάλεια για τους βιομηχανικούς φορείς προστατεύοντας τους ευαίσθητους πληθυσμούς, τους ευάλωτους πληθυσμούς. Αυτό θα μπορούσε κατά την άποψή μας να ενδυναμώσει την έκθεση που εν τέλει επεξεργάζεται η Επιτροπή Περιβάλλοντος. Ευχαριστώ. Συνάδελφος Ευχαριστώ κύριε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Για τα θέματα αυτά θέλω να ευχαριστήσω τη συνεισφορά του κύριου εισηγητή και να σας πω ότι κατανοώ γενικά και υποστηρίζω την πρόταση της Κομισιόν, αλλά έχω και ορισμένε αμφιβολίες. Συμφωνώ με τον εισηγητή για ορισμένε από αυτές τις αμφιβολίες και θεωρώ ότι χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο για να διευκρινιστούν αυτά τα θέματα. Έχω κάποιες αμφιβολίες ιδίω για τα τρόφιμα χωρίς γλουτένη. Η πρόταση αυτή είναι χρήσιμη, απαραίτητη, αντιμετωπίζει την εξέλιξη στην αγορά των τροφίμων, όπου υπάρχει και μια βαθμία αλλαγή του ρυθμιστικού πλαισίου και υπάρχουν και διαφορετικές βέβαια πρακτικές εφαρμογής στα κράτη-μέλη. Γι' αυτό είναι απαραίτητο να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε ορισμένες αντιμετωπίσεις οι οποίες περιορίζουν συγκεκριμένες κατηγορίες ε, τροφίμων. Είναι απαραίτητο λοιπόν να υπάρξει μια εναρμόνιση της ρυθμιστικής και κανονιστικής διαδικασίας στα κράτη-μέλη με την απλοποίηση των διαδικασιών για τις βιομηχανίες και ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πρέπει με τον τρόπο αυτό να εξασφαλίσουμε μια απλοποίηση η οποία όμως θα εξασφαλίσει και αντίστοιχο επίπεδο προστασία των καταναλωτών η, δεν πρέπει να θυγεί η πρόσβαση ειδικών κατηγοριών του πληθυσμού στα τρόφιμα αυτά. Δεν πρέπει όμω να χάσουμε από τα μάτια μα και την ανάγκη να υπάρξει μεγαλύτερο ανταγωνισμό, μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα και απλοποίηση σε κανονιστικό επίπεδο. Εμεί συμφωνούμε λοιπόν ιδιαίτερα με τον εισηγητή. Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει ακόμα αυτή η διαμάχη σε σχέση με τα προϊόντα χωρί γλουτένι τα οποία που θα πρέπει να διευκρινιστεί περισσότερο. Για τον κανονισμό 2041-2009, ο οποίο θα αντικατασταθεί από την, τροπο, από την νομοθεσία αυτή. Κινδυνεύουμε να βρεθούμε σε μια δύσκολη κατάσταση μέχρι την έγκριση του νέου κανονισμού. Γι' αυτό εγώ παρουσιάζω. Προτείνω να παραπέμψουμε όλες αυτές τις περιπτώσεις για τα προϊόντα χωρίς γλουτένη, παραδείγματος χάρη, στον κανονισμό ο οποίος προβλέπει την κοινοποίηση για τα στοιχεία αυτά. Θέλω να θέσω και δύο ερωτήματα στην Κομισιόν για το ζήτημα αυτό. Θα μπορούσε η Κομισιόν να μας διευκρινίσει αν αυτή η τροποποίηση που προτείνει τώρα στον κανονισμό είναι πρόσθετο κόστος για... Σημαίνει πρόσθετο πρέπει να υπομισθούν οι μικρομεσαίε επιχειρήσει, οι οποίε εργάζονται στον τροφιμικό τομέα και επομένω θα αποτελέσει μια, ένα πρόσκομα στην πρόσβαση αυτών των εταιριών και ένα βάρο για του καταναλωτέ. Δεύτερον θα μπορούσε η Κομισιόν να μα διευκρινίσει αν οι πολίτες που έχουν ειδικέ δυσανεξίε και προβλήματα, ιδίως αυτούς που χρειάζονται τρόφιμα χωρίς γλουτένη θα προστατευτούν, θα συνεχίσουν να προστατεύονται επαρκώς ω καταναλωτές που υπέχουν κινδύνους. Εάν δεν είναι θετική αυτή η απάντηση της Κομισιόν, ε, ενισχύονται οι αμφιβολίες που έχω και εγώ όπως ο εισηγητής και επομένως είναι απαραίτητο να επιληθούν τα θέματα αυτά το χειρότερο δυνατό. Η κυρία Τόγια. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω στους συναδέλφους από όλες τις πολιτικές ομάδες ότι συμφωνώ απόλυτα με την τοποθέτηση που δίνεται εδώ. Ο καθένας μας θέλει να καταλάβει περισσότερο κατά πόσο σωστή στόχη ή στόχη, η απλοποίηση και η έγκριση σωστή των προϊόντων ώστε να ικανοποιούνται όλες οι απαιτήσει των αγορών σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες ε, πηγαίνουν προς τη σωστή κατεύθυνση με αυτόν τον κανονισμό. Επίσης εκτιμώ πάρα πολύ που εμείς εδώ ε, καθώς και η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς γνωρίζουμε τις προσεγγίσεις και τους στόχους αλλά συνεχίζουμε να ξέρουμε ότι όσο πιο προηγμένη είναι η εσωτερική αγορά η ενιαία αγορά και η βιομηχανία όσο περισσότερες απαιτήσεις υπάρχουν για την ευημερία των πολιτών θα δημιουργηθεί καλύτερη βιομηχανία και καλύτερη εσωτερική αγορά και έτσι θα ικανοποιηθούν όλοι οι καταναλωτές. Ήθελα να εμβαθύνουμε όχι μόνο στην, στην Επιτροπή σήμερα, όχι μόνο στην Κομισιόν αλλά και μεταξύ μας θα πρέπει να υπάρχει λόγος απλοποίησης εφόσον ε, ελαττώνουμε το κείμενο σε σχέση με ορισμένους τύπους ευάλωτων πληθυσμών θα πρέπει να ξέρουμε γιατί το κάνουμε. Εδώ μιλάμε για βρέφη, για μικρά παιδιά, τρόφιμα για ειδικού ιατρικούς σκοπούς αλλά αφήνουμε απροστάτευτες τις κατηγορίες, ε, χωρίς αυτή την εγγύηση, ορισμένες κατηγορίες πληθυσμού που αποφεύγουν ε, τις ασθένειες χάρη σε, μια, σε ένα συγκεκριμένο τύπο διατροφής. Για αυτούς ε, ο τρόπος διατροφής είναι η μόνη θεραπεία που υπάρχει. Δεν είναι η ιατρική θεραπεία, αλλά είναι ο μόνος τρόπος ώστε να μην αρρωστήσουν. και ε, τους υποστηρίζουμε πλέον μόνο με απλές ε, συμβουλές, ε, ότι μπορούν να λάβουν μόνο συμβουλές που φυσικά βοηθούν εφόσον όμως οι άλλοι τις ακολουθήσουν γιατί είναι προαιρετικές. Εδώ μιλάμε για ζητήματα που δεν έχουν μόνο για μία, σχέση με μία υγιή ζωή, με μία καλή ζωή, έχουν σχέση με το να μην αρρωστήσει κάποιος. Εφόσον λοιπόν αποκλείουμε ορισμένες τέτοιες κατηγορίες ε, ε, συμμερίζομαι με την προσοχή που δίνουμε στα νέα διαιτητικά προϊόντα κατά και τα κτλ. Πρέπει να προσφέρουμε όλο και περισσότερες εγγυήσει και όχι να αφήσουμε τους καταναλωτές, τους πολίτες ε, στα χέρια μιας συμφεροντολόγου διαφήμισης κατά κάποιο τρόπο. Εμείς και μέσω ανεξάρτητων αρχών και μέσω μιας επιστημονικής αξιολόγησης όλο και πιο βαθιάς πρέπει να προσφέρουμε αυτές τις διασφαλίσεις με την ομοθεσία μας. Εφόσον εμείς διασφαλίσουμε αυτά τα επίπεδα διατροφικής ασφάλειας, βοηθάμε επίσης και την καινοτομία στις επιχειρήσεις, επειδή σήμερα υπάρχει ένας ολόκληρος τομέας διατροφικής τεχνολογίας που θα επιτρέψει στις βιομηχανίες μας να αυξήσουν τις τεχνολογικές τους ικανότητες και την προσαρμογή τους. Και αυτή είναι η βιομηχανική καινοτομία που μας θέτει στο προσκήνιο και που επίσης αφορά την υγεία των πολιτών και χαμηλότερα κόστη όσον αφορά τη θεραπεία ε, ασθενειών. Αφορά λοιπόν την υγεία, τη βιομηχανία και τον προπολογισμό όλο αυτό το ζήτημα. Εγώ πιστεύω ότι αυτή η λύση είναι χειρότερη για, ορισμένους τρο για ορισμένες ασθένειες ε, οι οποίες εξαρτώνται από τη σωστή διατροφή. Εγώ πιστεύω ότι εδώ μιλάμε για επιδείνωση. Πιστεύω ότι οι αμφιβολίες που διατύπωσαν πολλοί και εδώ και στις υπόλοιπες ε, επιτροπές ε, θα βρουν κάποια ανταπόκριση μέσω τροπολογιών. Θα πρέπει να κάνουμε κάτι για όλες αυτές τις πτυχές, ε, διατηρώντας φυσικά ταυτόχρονα, δεν χρειάζεται να παραβλέψουμε την απλούστευση και τα προφίλ διατροφής και όλα αυτά. Ωστόσο δεν πρέπει να αφήσουμε απροστάτευτες κάποιες κατηγορίες. Ε, Σύμφωνο με αυτό που είπατε ότι για τα παιδιά ας πούμε ε, πρέπει να προσφέρουμε τη διασφάλιση. Δεν πρέπει να επιδεινώσουμε την νομοθεσία για να απλοποιήσουμε την αγορά. Πρέπει να βοηθήσουμε στην ανάπτυξη της αγοράς και των βιομηχανιών και της τεχνολογίας βελτιώνοντας την ποιότητα για τους καταναλωτές. Στο στάδιο αυτό της συζήτησης θέλω να σταθώ μονάχα σε ένα σημείο. Και άλλοι συναδελφοί το έχουν θίξει το σημείο αυτό, αλλά θα πρέπει να επιμείνουμε ίσως. Θέλω να επιστήσω την προσοχή σας στα προβλήματα τα οποία μπορούν να προκύψουν από την τροποποίηση των συνδικών διανομής των τροφίμων χωρίς γλουτένη η δυσανεξία στη γλουτένη είναι πολύ διαδεδομένη. Περίπου 1% του πληθυσμού καλύπτει αυτή η δυσανεξία. Τα θύματα αλλεργίας στη γλουτένη είναι όλο και περισσότερα, είναι αντισυγητική αύξηση των, του αριθμού των θυμάτων και η διάγνωση αυτής της ασθένειας είναι πολλές φορές πολύ δύσκολη. Η μόνη θεραπεία που προβλέπεται για τους ασθενείς είναι η διατήρηση μιας δίαιτας χωρίς γλουτένη. Οποιαδήποτε τώρα απόκληση από αυτήν την δίαιτα δημιουργεί προβλήματα κινδύνου ε, καρκίνου του παχαιοσεντέρου, προβλημάτων στο, στα οστά και άλλες αυτοάνωσες ασθένειες. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τα τρόφιμα που έχουν σε στόχο ειδικέ ιατρικέ δίαιτες, αν ακολουθήσουμε αυτά που μα προτείνει η Κομισιόν, η τροποποίηση αυτή μπορεί να τροποποιήσει και την εκετοθεσία των προϊόντων χωρί γλουτέν και να κάνει πιο δύσκολη για του ασθενεί την ανάγνωση τη σύσταση αυτών των φαρμακών. Κάποιε χώρε όπω η Ιταλία, η Αυστρία, η Γερμανία και κάποιε άλλε έχουν ήδη τονίσει την αντίθεσή του σε μια τέτοια τροποποίηση η οποία θα οδηγήσει σε αθέλητα σφάλματα ασθενών και θανάσιμα κιόλα, που θα έχουν αρνητικά αποτελέσματα για την υγεία του. Έχω καταθέσει όπως και άλλοι τροπολογίες για να διατηρηθεί η επαρκής ορατότητα και η ασφάλεια των προϊόντων αυτών χωρίς γλουτένη που είναι απαραίτητα για να μπορέσουμε να αποφύγουμε βαριές επιπλοκές για αυτούς οι οποίοι έχουν ασθένειες αυτού του είδου και επομένως ελπίζω ότι αυτές οι τροπολογίες θα υποεστηριχθούν. Σας ευχαριστώ. Κομισιόν. Ευχαριστώ. Κομισιόν θέλει να συμπληρώσει κάτι. Παρακαλώ. Έχετε το λόγο. Ναι, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ναι, πράγματι έθεσαν κάποιες ερωτήσεις προς την Κομισιόν Τι οποίες θα ήθελα να απαντήσω. Πρώτα απ' όλα όμως θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την έκθεσή του. Νομίζω πως ε, το γεγονός πως αναγνωρίζεται η απαραίτητη όθηση της Κομισιόν είναι ικανοποιητικό. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τους υπόλοιπους βουλευτές ε, που παρενέβησαν και θα ήθελα να προσπαθήσω να απαντήσω σε κάποιες από τις ανησυχίες τους. και να προσπαθήσω να καθησυχάσω, να καθησυχάσω κάποιους φόβους για, τους, ε, για τα κενά που θεωρούν ότι παρουσιάζει η πρόταση. Οι ανησυχίες που ακούσαμε σήμερα οφείλονται ίσως σε πληροφορίες που ελήφθησαν από τη μία πλευρά των ενδιαφερομένων γιατί δεν λέω πως ε, άλλα ενδιαφερόμενα μέρη πως οι καταναλωτές ε, υποστηρίζουν πλήρως την πρόταση και αυτό είναι σημαντικό γιατί την ανέλησαν εις βάθος. καταναλωτέ, οι οποίοι έχουν, ε, έχουμε τη γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Γραφείου των Ενώσεων Καταναλωτών ε, βασική ε, συνομοσπονδία οργανώσεων καταναλωτών που προσωπεί τα συμφέροντά τους σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. υπονοήθηκε πως οι κανόνες ε, υποχωρούν εδώ πέρα. Δεν ισχύει αυτό γιατί η πρόταση είναι αποτέλεσμα της εξέλιξης της νομοθεσίας ε, σε πιο οριζόντιους τομείς ε, όπως η νομοθεσία για τα συμπληρώματα τροφίμων, για τα πρόσθετα και μεταλλικά στοιχεία τροφίμων, διάφορες άλλες ουσίες. Περισσότερο από οτιδήποτε άλλο λοιπόν και βεβαίως ε, αποτέλεσμα του κανονισμού για τις προσφυγές, ο οποίος συζητήθηκε στο Κοινοβούλιο και πιο πρόσφατη νομοθεσία, η υιοθέτηση του κανονισμού για την πληροφόρηση των καταναλωτών ε, για τα τρόφιμα. Ξεκινώντας λοιπόν από το ζήτημα που ε, προκάλεσε τις περισσότερες ανησυχίες, τα προϊόντα χωρίς γλουτένη, δεν ξέρω από πού προκύπτει η ιδέα πως οι κανόνες μειώνουν ε, την προστασία των καταναλωτών. Αλλά μπορώ να διαβεβαιώσω τα μέλη της Επιτροπής πως ε, δεν ε, ισχύει αυτό, όπως δεν υπάρχει και επιπλέον κόστος που θα επιβληθεί. τι συμβαίνει με τον κανονισμό περί τροφίμων χωρίς γλουτένης. Το μόνο το οποίο έχουμε είναι απαιτήσει σήμανσης για το πότε η δήλωση χωρίς γλουτένη ή με χαμηλή γλουτένη μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Και σας διαβεβαιώ πως αυτό το οποίο προτείνει η Κομισιόν είναι να έχουμε ακριβώς την ίδια διατύπωση των διατάξεων που ισχύουν εκεί και να τις μεταφέρουμε. Ενώ αρχικά είχαμε υποβάλει την πρόταση πως θα πρέπει να γίνει ναι, σύμφωνα με τον κανονισμό περί προσφυγών, αλλά από όταν ευθύθηκε ο κανονισμός ε, πληροφόρηση ε, των καταναλωτών για το τρόφιμα θεωρήσαμε πως ήταν προσφορότερο. Οπότε σας διαβεβαιώ πως δεν θα αλλάξει τίποτα όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών, όσον αφορά το κόστος των ε, χρηστών και των εταιριών. Η κυρία Γκροστέτ έθεσε έμφαση στη συζήτηση περί προϊόντων αδυνατίσματος. Γνωρίζετε πως το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο το 2006 ενέκριναν τον σχετικό κανονισμό όπου αναφέρεται πως ε, οι ισχυρισμοί ε, τροφίμων ε, περί αδυνατίσματος κτλ ήταν αποδεκτά. Ήταν αποδεκτή, με Και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε αυτό, όπως επίσης να αντιμετωπίσουμε και το γεγονό πως ε, τέτοιοι ισχυρισμοί είχαν γνωστοποιηθεί στην Κομισιόν, αξιολογήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων, οπότε ξέρετε πως ε, ασφάλεια εφίσταται και σας διαβεβαιώ πω η όροι χρήσης ε, τέτοιων ε, ισχυρισμών είναι ακριβώς ε, αυτοί που υπάρχουν στην υφιστάμενη οδηγία, η 98-6 δηλαδή. Αυτό το οποίο κάναμε άρα είναι να έχουμε μια θετική ψήφο για τους ισχυρισμούς αυτούς που έχουν εγκριθεί και αυτοί αφορούν και τα υποκατάστατα γάλακτος συγχωρείτε, τροφίμων, ε, γευμάτων. Ακούσαμε επίσης κάποιες ανησυχίες για προϊόντα τα οποία πολλούνται ως ε, προϊόντα τα οποία αντικαθιστούν μια ε, πλήρη καθημερινή διατροφή. Δεν μιλάμε δηλαδή για κάποιες μπάρες που αντικαθιστούν ένα γεύμα, αλλά ε, προϊόντα τα οποία αντικαθιστούν ολόκληρη την καθημερινή διατροφή. Και μεταξύ αυτών υπάρχουν και τα προϊόντα εκείνα τα οποία έχουν ε, πολύ λίγες θερμίδες, μεταξύ 400 και 800 κιλοκάλ. Οπότε ακούσαμε και τα κρατη και το Κοινοβούλιο πως όσον αφορά τα, αυτά τα προϊόντα μπορεί να υπάρχουν κάποιες ανησυχίες και η Κομισιόν βεβαίως ε, μπορεί να συζητήσει κάποιες αλλαγές, στην πρότασή της όσον αφορά αυτά τα συγκεκριμένα προϊόντα. Όμως δεν ε, θεωρούμε πως ε, τρόφιμα για αθλητές είναι το ίδιο προϊόν. Οι αθλητές δεν είναι ευάλωτοι θα έλεγα και η εμπειρία έχει δείξει πως όλα αυτά τα χρόνια που είχαμε την δυνατότητα να ορίσουμε κανόνες για τα τρόφιμα για αθλητές και για συγκεκριμένες κατηγορίες δεν ε, μπορέσαμε να το κάνουμε γιατί είτε τα επιστημονικά στοιχεία άλλαζαν συνεχώς και άρα ο φόβος ε, του να σταματήσουμε την καινοτομία ήταν τόσο μεγάλος ώστε και οι ίδιες οι εταιρείες δεν ήθελαν να έχουμε έναν συγκεκριμένο κανόνα. Και να πω επίσης πως στον πρόσφατο κατάλογο ισχυρισμών ε, που εγκρίθηκαν από την μόνιμη επιτροπή και θα χρειαστεί να εξετάσετε προσεχώς υπάρχουν δύο-τρεις ισχυρισμοί όσον αφορά τους αθλητές οπότε η πρότασή μας νομίζω λειτουργεί και η δουλειά απόδειξη όσον αφορά τις τσίχλες ε, βεβαίω να σας ακούσουμε κυρία Γκροστέτ αλλά πρέπει να αντιδράσω σε αυτό το οποίο είπατε ότι δηλαδή ε, χρειαζόμαστε αυτά τα γάλατα ε, Ανάπτυξη γιατί πρέπει να προστατεύσουμε τα παιδιά από διάφορα ζυζανιοκτώνα που μπορεί να περιέχουν αυτά. Αυτό είναι προσβολή θα έλεγα για τη βιομηχανία του γάλακτος γιατί αν τους πείτε πω τα προϊόντα τους λόγω διαφόρων ζυζανιοκτώνων δεν είναι κατάλληλα για παιδιά μεταξύ ενός και τριών ετών νομίζω πως θα υπάρξει εξέγερση από τη βιομηχανία. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στα επιχειρήματα που χρησιμοποιούμε για να πούμε κάτι. Επιπλέον, ε, είμαστε διατεθειμένοι να εξετάσουμε κάτι ε, όσον αφορά την καινοτομία και να διευκολύνουμε την καινοτομία. Τώρα, όσον αφορά την ανεξάρτητη αξιολόγηση, θεωρώ πως η αξιολόγηση της ΕΦΣΑ είναι ανεξάρτητη, δεν έχω καμία αμφιβολία. Ο χρόνος μου έχει τελειώσει, αντιλαμβάνομαι, οπότε θα σταματήσω εδώ. Ευχαριστώ. Frau Grostet Γκροστέτ ήθελε να λάβει ξανά τον λόγο. Σύντομα. Ναι κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ που μου δίνετε για λίγο το λόγο. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Δεν συμφωνώ με όσα είπε συστηματικά ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ναι, ο κανονισμός για τους ισχυρισμούς είναι ένας κανονισμός που τον γνωρίζω καλά, τον έχω δουλέψει όσον αφορά τον κανονισμό για την ενημέρωση των καταναλωτών. Τον γνωρίζω επίση καλά το θέμα είναι ότι αυτοί οι κανονισμοί δεν ισχύουν αυτή τη στιγμή, δεν ισχύουν ακόμη. Διότι ο κανονισμός για τους ισχυρισμού ψηφίστηκε πρόσφατα, κύριε εκπρόσωπε της Κομισιόν, δεν ισχύει ακόμα δεν έχουμε κρατήσει δεν έχουμε την απαραίτητη πείρα για να ξέρουμε κατά πόσο θα είναι επαρκώς θετικά και στις συνέπειες για την προστασία των καταναλωτών αλλά και ταυτόχρονα για την προστασία της αγροδιατροφικής βιομηχανίας η οποία χρειάζεται αυστηρά πλαίσια για να γνωρίζει προς τα ποδεύει. Δεν συμφωνώ λοιπόν με αυτό. Γι' αυτό το λόγο σας ζητάμε να συμπεριλάβετε στην πρότασή σας το γάλα για μικρά παιδιά ενό έω τριών ετών, επειδή γνωρίζουμε πολύ καλά ότι είναι πιο ευαίσθητα αυτά τα μικρά παιδιά, πιο ευάλωτα και ότι χρειάζονται γαλακτοκομικά προϊόντα με λιγότερη περιεκτικότητα σε ζενιοκτώνα. Γνωρίζετε, έχουμε κανονισμό για τα ζενιοκτώνα. Ξέρετε ότι πρέπει να τα προφυλάξουμε αυτά τα παιδιά ενό έω τριών ετών. Το ίδιο ισχύει για τα άτομα με δυσανεξία στη γλουτένη στη λακτόζη. Χρειαζόμαστε να υπάρχει κάποια αυστηρότητα. Η αγροδιατροφική βιομηχανία επίσης χρειάζεται να γνωρίζει τι πρέπει να πράξει. Ο κανονισμός για τους ισχυρισμού και ο κανονισμός για την ενημέρωση των καταναλωτών δεν επαρκούν σήμερα. Χρειαζόμαστε κάποια περισσότερη πείρα. Θα το δούμε σε 3, 4, 5 χρόνια. Αλλά προς το παρόν δεν έχουμε το περιθώριο να παραβλέψουμε, ας το πω έτσι, αυτούς τους πληθυσμούς που χρειάζονται συγκεκριμένα τρόφιμα. Σας ευχαριστώ. Κύριε Τάκκουλα, θέλετε να πείτε κάτι παραπάνω, να προσθέσετε κάτι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. σε σχέση με αυτά που είπε η κυρία Γκροστέτ εν κατακλείδη. Ναι, είναι σωστό αυτό που λέει. Όπως είπα όπως και εγώ στην αρχή της παρέμβασής μου, εμείς είμαστε συντάκτες γνωμοδότησης. Η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή είναι η Επιτροπή Περιβάλλοντος. Εκεί θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι θα γίνουν πιο σαφείς αυτές οι διατάξεις. Από τη δική μας πλευρά, εμείς θέλουμε να τονίσουμε την ανάγκη να υπάρχει σαφέστερη προστασία του καταναλωτή μέσω της καλύτερης παροχής πληροφοριών. Το θέμα της ε, δυσανεξίας στη γλουτένη, αυτό είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα, ένα μεγάλο ερώτημα όπως ανέφερε και η Κομισιόν στην έκθεση ΡΙΙΣ, αναφέρεται, αναφέρθηκε μάλλον, ότι οι διατάξεις για την ε, γλουτένη ή την ε, λακτόζη και τη δυσανεξία σε αυτά τα προϊόντα να αντιμετωπιστούν πιο ενδελεχώς σε άλλα νομοθετήματα. Εγώ πιστεύω όμως θα ήταν χρήσιμο να ήταν όλα σε ένα έγγραφο και αυτό θα έκανε πιο σαφή την κατάσταση. Ώστε ο καταναλωτής να γνωρίζει πάντα τι τρώει. Για τη δική μας πολιτική ομάδα είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε τι γίνεται σε επίπεδο ερευνητικό σε σχέση με τα προϊόντα αυτά και να ξέρουμε όλοι τι περιέχουν τα προϊόντα αυτά. Η σημερινή συζήτηση κατέδειξε ότι δεν μπορεί μια εταιρεία να κάνει σχισμούς για τα προϊόντα της που δεν στέκονται. Χρειάζονται λοιπόν αυτά να προσδιοριστούν καλύτερα. Υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι λένε τις Παναγιά στα μάτια για τα τρόφιμα τα οποία παράγουν, αλλά αυτά δεν έχουν καμία πραγματική βάση. Γι' αυτό το λόγο είναι απαραίτητο να εξασφαλίσουμε την προστασία του καταναλωτή. Αυτά λοιπόν κύριε Πρόεδρε, αυτά ήθελα να πω εγώ. Νομίζω ότι ήταν πολύ θετική η συζήτηση και όπως είπα θα πρέπει να επανέλθουμε στο θέμα του τι θα προσθεθεί ως τροπολογία στο κείμενο. Έχουμε καιρό, όπως σας είπα, μέχρι την Τρίτη για την κατάθεση τροπολογιών και με τον τρόπο αυτό μπορούμε να βοηθήσουμε και την Επιτροπή Περιβάλλοντος, που είναι η αρμόδια, αλλά εγώ, όπως σας είπα, εστίασα στα θέματα που είναι στις δικές μας αρμοδιότητες. Ευχαριστώ πολύ, λέω πρόεδρος. 17 Ιανουαρίου είναι η τελική προθεσμία για τις τροπολογίες. Έχει επιληθεί και αυτό το σημείο, λοιπόν. 23, 24, 25 Ιανουαρίου είναι η επόμενη μας συνεδρίαση και να σας πω και το εξής. Στις 23 Ιανουαρίου θα γίνει η συγκρότηση της Επιτροπής μας με την εκλογή Προέδρων κτλ. 23, όχι στο Στρασβούργο, στις Βρυξέλλες, 23 Ιανουαρίου. Σας ευχαριστώ τα μάλα και σας εύχομαι καλή συνέχεια.